Η συνεδρίαση ε, θα αναμεταδίδεται μέσω διαδικτύου. Να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Σας έχει διανημηθεί η ημερήσια διάταξη από τις 8 Μαρτίου, οπότε δεν μπορεί, θα την έχετε λάβει. Έχω ένα αίτημα από τον κύριο Χέφνερ να προσθέσουμε στην ημερήσια διάταξη την εξέταση για την ερμηνεία του άρθρου 128 του κανονισμού, θέμα για το οποίο είμαι εγώ Το αίτημα λοιπόν του κυρίου Χέφνερ να συζητήσουμε στη σημερινή συνεδρίαση την ερμηνεία του άρθρου 128 του κανονισμού ε, νομίζω ότι μπορούμε συγχωρείτε, υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, δεν ακούμε τον Πρόεδρο. Si τώρα. Λοιπόν, ο συνάδελφος Γκουαλτιέρη, ο οποίος είναι σκιώδης εισηγητής για την έκθεση του συναδέλφου Άντριου Νταφ για την ε, εκλογική νομοθεσία, δεν μπορεί να παραστεί σήμερα και ζητά να κάνουμε αύριο το πρωί τη συζήτηση επί του θέματος αυτού. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, μπορούμε να τροποποιήσουμε την ημερήσια διάταξη. Αυτό μας επιτρέπει να ελπίσουμε να ολοκληρώσουμε νωρίς και επομένως να γίνει σήμερα η συνεδρία των συντονιστών και όχι αύριο το πρωί και αύριο το πρωί κατά τι ώρες που προβλεπόταν η συνεδρία των συντονιστών, 9 με 10, ε, μπορούμε να βάλουμε την έκθεση DAF, στις 9 το πρωί λοιπόν. Συνοψίζω λοιπόν, Αύριο το πρωί θα συμπεριλάβουμε την έκθεσή μου για την ερμηνεία του άρθρου 128 του κανονισμού, όπως ζήτησε ο συνάδελφος Χέφνερ. Αφαιρείται από τη σημερινή συνεδρίαση η συζήτηση για την έκθεση DAF που ήταν στο σημείο παριθμών 6 της ημερησίας διάταξης και θα το συζητήσουμε αύριο το πρωί. Το είχαμε χωρίσει σε δύο τμήματα, μία γενική συζήτηση για τις τροπολογίες και ψηφοφορία. Ε, αύριο το πρωί στις 9 θα γίνει όλη η συζήτηση. Σήμερα το, πρωί, σήμερα το απόγευμα, συγγνώμη, στο τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, γύρω στις 5.30, την ε, συνεδρίαση των συντονιστών, ελπίζω. Όσον αφορά τη συνεδρίαση των συντονιστών, έχω λάβει ένα μήνυμα από τον συνάδελφο Ταρκόφσκι, ο οποίο είχε ζητήσει να μείνει για αύριο το πρωί η συνεδρίαση των συντονιστών, γιατί στη συνεδρίαση αυτή θα πρέπει να συζητήσουμε και την επίσκεψή μα στην Πολωνία και φυσικά ο κύριο Ταρκόφσκι έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο για την επίσκεψη αυτή. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε κάλλιστα όλα τα υπόλοιπα και αύριο να μιλήσουμε για την επίσκεψη στην Πολωνία. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις, τα ρυθμίσουμε έτσι. Ο κύριος Νταφ. Δεν ε, ε, έχω κάποια ένσταση καταρχήν. Θα ήθελα όμως να ζητήσω το εξής. Χρειαζόμαστε τον κατάλληλο χώρο και χρόνο για να συζητήσουμε το θέμα της μεταρρύθμισης εκλογικής ε, διαδικασίας επί της ουσίας. Ε, άρα τώρα να το στριμώξουμε μαζί με τη συνεδρία των συντονιστών αύριο το πρωί και να έχουμε τον Επίτροπο Σεύκοβιτς ε, στο τέλος του πρωινού, νομίζω ότι θα μεταράξει Uh, my request is I... Άρα... Προτείνω να ε, τηλεφωνήσουμε στον Επίτροπο τόσο ώστε να καταφτάσει στις 11 και 4 αύριο το πρωί ούτως ώστε να ε, έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο στη διάθεσή μας για να συζητήσουμε την έκθεσή μου. Ούτως ή άλλως τις τριμώχνουν πάντα την έκθεσή μου στην μερίσια διάταξη της Επιτροπής. Ζητώ συγγνώμη κύριε Νταφ. Ίσως δεν να κατανοητός. Η πρότασή μου ήταν να γίνει συνεδρίαση των συντονιστών απόψε, στο τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, προκειμένου να έχουμε περισσότερο χρόνο αύριο και να τον αφιερώσουμε όλο στην εκθεσή σα. Δηλαδή, θα γίνει απόψε συνεδρία των συντονιστών και η συνεδρίαση θα ξεκινήσει αύριο το πρωί στις 9 και θα έχουμε έτσι εξασφαλίσει χρόνο ε, που είχαμε για τη συνεδρίαση των συντονιστών αύριο το πρωί. Έχουμε χρόνο λοιπόν. Το δέχεστε κύριε Ντάφ. Yes, okay. Um, Μάλιστα. Αλλά θα ήθελα να ζητήσω να αρχίσουμε ακριβώς στις 9 αύριο το πρωί. E Εγώ εδώ θα είμαι, να πούμε και στους άλλους να έρθουν. Ε, ε βλέπω όλοι να χνεύουν καταφατικά. Ας φροντίσουμε λοιπόν να είμαστε όλοι εδώ στις 9. Θέλει και ο κύριο Σούλτ το λόγο για το σημείο αυτό. Ο κύριο Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι βεβαίω πω είναι δύσκολο να συντονίζουμε τα προγράμματα όλων των βουλευτών γιατί ο καθένας πρέπει να είναι κάπου αλλού παρόν. Να υπενθυμίσω πως και εγώ είμαι σκιώδης συγητής στην έκθεση του κυρίου Νταφ και δυστυχώς ε, έχουμε αύριο το πρωί συνεδρίαση της Επιτροπής ΙΝΤΕ. Οπότε πρέπει να τηρήσουμε και το αρχικό πρόγραμμα για να μπορούμε να προγραμματίσουμε και το τι θα, θα κάνουμε. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να συμμετάσχουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν να το λάβετε υπόψη για το μελλοντικό προγραμματισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς ε, προσπαθώ να τους ε, έχω ευχαριστημένους όλους και σήμερα ειδικά μέχρι τελευταία στιγμή καθόμαστε και προσπαθούσαμε να αλλάξουμε τη σειρά τη ημερήσιας διάταξης για να τους έχουμε όλους ευχαριστημένους. Σας παρακαλώ λοιπόν κύριε Σόλτς να έχετε υπομονή αυτή τη φορά. Ε, λαμβάνω υπόψη τη σύστασή σα ε, ως υπόδειξη για το μέλλον, αλλά σα παρακαλώ μην μου ζητήσετε να αλλάξω πάλι την ημερήσια διάταξη, διότι πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δεν έχω άλλε ανακοινώσει του Προέδρου. Πρέπει όμω να εγκρίνουμε τα πρακτικά τη συνεδρίαση τη 31η Ιανουαρίου και 1η Φεβρουαρίου του 2011, τη 7η Φεβρουαρίου, τη 14η Φεβρουαρίου και τη 17η Φεβρουαρίου. Είναι διαθέσιμα τα πρακτικά. Αν δεν γίνουν παρατηρήσει μέχρι το τέλο τη συνεδρία, θεωρούνται ω εγκριθέντα. Και μπορούμε να περάσουμε πλέον στα σημεία 4 και 5, για τα οποία είναι εισηγητή ο υποφαινόμενος και θα ήθελα να σας παρουσιάσω από κοινού. Διότι όπως ε, γνωρίζετε η διοργανική συμφωνία σχετικά με ένα κοινό μητρό διαφάνειας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή μα. Και κατά συνέπεια θα πρέπει να προτείνουμε και κάποιες ε, τροποποίησεις για τον κανονισμό, οι οποίες απορρέουν από την έγκριση της συμφωνίας. Όσον αφορά τη συμφωνία, θα πρέπει είτε να τη δεχτούμε είτε να την απορρίψουμε. Δεν μπορούμε να την τροποποιήσουμε. Επί του κανονισμού, προφανώς, ε, υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε και τροποποίησεις. Θα ήθελα όμως να συζητήσουμε από κοινού τα δύο θέματα, γιατί ουσιαστικά ένα θέμα είναι. Το έχουμε συζητήσει το θέμα της συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου στη συνεδρίαση της 1ης Φεβρουαρίου όταν είχε έρθει και η Αντιπρόεδρος Γόλης εδώ και μας είχε παρουσιάσει το περιεχόμενο της ε, διοργανικής αυτής συμφωνίας για ένα μητρό, το οποίο δεν θα λέγεται πλέον μητρό εκπροσώπων συμφερόντων, αλλά μητρό διαφάνειας. Η καινοτομία έγκυται στο γεγονός ότι πλέον πρόκειται για ένα κοινό μητρό μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου και μάλιστα είμαστε εν αναμονή και τα πράγματα είναι πολλά υποσχόμενα και τη συμμετοχή του Συμβουλίου. Δηλαδή το Μητρό θα είναι κοινό και για τους ε, ε, ε Θα μας πει και ο Επίτροπος Εύκοβιτς αύριο τι ε, ε συμβαίνει αλλά θα δούμε αν μπορούμε να έχουμε ένα κοινό μητρό της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για το πρώτο σημείο τώρα τι άλλο να σας πω. Αν θυμάμαι καλά, το πρόβλημα του Μητρώου Διαφάνειας για τους εκπροσώπους συμφερόντων είχε ήδη τεθεί από την έκθεση ΣΤΑΜΠ στην προηγούμενη νομοθεσία, η θετία, το 2008 και τότε υπήρχε υποστήριξη από τα μέλη της Επιτροπής. Η έκθεση είχε και μια ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου, η οποία θα ήταν υπεύθυνη για την εκπόνηση αυτής της ε, συμφωνίας. Συστάθηκε η ομάδα. Η πρόεδρος της ομάδας ήταν η συνάδελφος Γουόλης, ε, συμμετείχα και εγώ, συμμετείχε και η κυρία Ισαμπέλ Τουράν και ο συνάδελφος Γιολάινεν και εργαστήκαμε προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτό το έγγραφο. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτού του εγγράφου αυτής της συμφωνίας. Η εγγραφή είναι δικαίωμα, δεν είναι υποχρέωση. Όποιο θέλει να απολαμβάνει συγκεκριμένων ε, πλεονεκτημάτων πρέπει να είναι εγγεγραμμένο σε αυτό το Μητρό και για να μπορέσει να εγγραφεί στο Μητρό θα πρέπει να δώσει και κάποιε πληροφορίε, κυρίω ε, οικονομική φύσεω, για ε, πιθανή συνεισφορά που λαμβάνει από πλευρά ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Δεν είναι υποχρεωμένο, αλλά εάν δεν εγγραφεί στο Μητρό δεν θα απολαμβάνει των δικαιωμάτων που απορρέουν από το Μητρό. Δεύτερον, το μητρό αυτό το είχαμε σκεφτεί ως ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο μητρό. Προβλέπεται λοιπόν και ένα τμήμα το οποίο δεν αφορά τους εμπορικούς φορείς αλλά τους μη εμπορικούς φορείς που μπορούν παρόλα αυτά να συνεισφέρουν στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα αλλά πρόκειται στον ίδιο κώδικα διοντολογία και του ίδιους κανόνες ουσιαστικά. Σας έχω ήδη πει ότι μεταξύ των βασικών υποχρεώσεων όσων θέλουν να εγγραφούν στο Μητρό θα πρέπει να δώσουν πληροφορίες για τη δομή του φορέα, ποιο είναι ο προέδρο ποια είναι τα όργανά του και κυρίως ε, οικονομικές πληροφορίε. Νομίζω ότι δεν ε, πρέπει να σας πω κάτι επιπλέον για τη συμφωνία αυτή. δεν μπορούμε να την τροποποιήσουμε όπως σας είπα, είναι ή το δεχόμαστε ή το απορρίπτουμε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το δεχτούμε διότι θεωρώ ότι πρόκειται για ένα ε, βήμα ε, προς την περαιτέρω διαφάνεια των θεσμικών οργάνων. Τώρα, οι τροποποίησεις που πρέπει να γίνουν στον κανονισμό. Οι τροποποίησεις που πρέπει να γίνουν στον κανονισμό είναι απαραίτητες και γίνονται ε, υπό την έννοια του άρθρου 127 θα έχουμε τροποποίηση στο άρθρο 9 που αφορούσε το παλιό μητρό προσώπων συμφορώντων και στο παράρτημα 10 που ήταν κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες ε, με βάση το άρθρο 9. Να σας πω ότι το νέο μητρό και ο κανονισμός βασίζεται στη δομή του προηγούμενου κανονισμού. Αυτό που έχει σημασία ε, είναι ότι το Κοινοβούλιο είναι αρμόδιο για μία σειρά από λεπτομέρειες. Η εγγραφή στο Μητρό είναι υποχρεωτική για όποιον θέλει να έχει πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά το Κοινοβούλιο είναι αρμόδιο για τους πιο διεξοδικούς κανόνες, να καθορίζει δηλαδή ποιες είναι οι προϋποθέσεις ε, ε, και κυρίως πόσο οργανώνονται όλοι όσοι ε, έχουν εγγραφεί στο Μητρό. Επιβεβαιώνεται εκ νέου λοιπόν και η ελευθερία των κοσμητόρων, η διαδικασία έκδοσης δελτίου ελευθέρας εισόδου, το πώς μπορεί να εφαρμόσει το κώδικα διοντολογίας ακόμα και σε αυτούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας και όλα αυτά στη συνέχεια ενσωματώνονται στο σημείο Β του παραρτήματος 10 πέρα από τις αλλαγές που γίνονται στο άρθρο 9. Προτείνεται το αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει τα μέτρα για την εφαρμογή του Μητρώου και της Συμφωνίας ε, να είναι το, το γραφείο της Προεδρίας κατόπιν προτάσεις του Γενικού Γραμματέα. Υπάρχουν επίσης και κάποιες ε, πιο λεπτομερείς ε, τροποποιήσεις, έχουν ομαδοποιηθεί κάποια στοιχεία στο άρθρο 9, καταργούνται οι διατάξεις οι οποίες δεν ισχύουν λόγω της νέας συμφωνίας, αλλά νομίζω ότι η τροποποίηση του κανονισμού μας ε, επιτρέπει να διατηρήσουμε τις βασικές μας αρμοδιότητες, δεν υπάρχουν προβλήματα, θα πρέπει να το εγκρίνουμε και δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά. Για να είμαι σαφής, ε, επί της ουσίας η εγγραφή στο Μητρό είναι υποχρεωτική για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να τους δώσει άδεια εισόδου. Αλλά δεν αποκλείονται οι υπόλοιπες αρμοδιότητες και εξουσίες ε, επί της οργάνωσης. Η συγγενείς, οι βοηθοί και όλοι αυτά μπορούν να έχουν πρόσβαση παρά το γεγονός ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό. Αυτό ούτως ή άλλως ισχύει ήδη και μένουν όσοι έχουν αυτά τα πράγματα, δεν αλλάζουν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση. Ε, δεν ξέρω ποιος θέλει το λόγο. Ο κύριος Κρέφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντικό αυτό το έγγραφο που θα εγκρίνουμε. Είναι δύο εκθέσεις. Μία για τον κανονισμό που θα αλλάξει αλλά και η πολιτική έκθεση. Και διαφάνεια είναι σημαντική. Καλό είναι ότι αλλάξαμε και το όνομα, το Μητρό Διαφάνειας. Δηλαδή καλό είναι όταν τα θεσμικά όργανα, τα κοινοβούλια είναι διάφανα. Τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν και πολύ υπέρα, αλλά τώρα το θεωρώ κάτι καλό, το μητρό των λόμπι. Όσον αφορά τώρα το Συμβούλιο και το κοινό μητρό με το Συμβούλιο, εκεί πέρα θα ήθελα πιο έντονη την διατύπωση. Γιατί θεωρώ πως οι πολίτες μας δεν κάνουν την διάκριση μεταξύ κομισιών, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ένα κοινό μητρό με λογική διατύπωση να μην υπάρχει πλέον χώρος ερμηνεών. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Ένα κοινό δημόσιο μητρό. Και αυτό είναι, το ότι είναι δημόσιο είναι θετικό ήδη. Ε, στην Κομισιόν μπορεί κανείς να δει με πόσα λεφτά επιδοτούνται αυτοί οι άνθρωποι. Και μπορώ να πω ήδη και σήμερα για το λέω πάντα δηλαδή και στους επισκέπτες, πως έχουμε και σήμερα ένα εθελοντικό μητρό, αλλά ε, είναι, θα πρέπει να είναι δεσμευτικό, ειδικά όσον αφορά το ε, Συμβούλιο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Επίσης θα πρέπει να ορίζετε πό, όταν παραδιάζονται κανόνες, ποιες είναι οι συνέπειες για να ξέρει ο καθένας πως υπάρχουν και συνέπειες όταν δεν τηρεί τους κανόνες που θέτουμε. Σε γενικές γραμμές είναι επιτυχημένη έκθεση και νομίζω πως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα δύο θεσμικά όργανα θα κάνουν ένα βήμα προς τα εμπρός γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ προκαταλήψεις για την Ευρώπη, πως εκεί πέρα είναι όλα διαφανή και τα λοιπά. Με το μητρό αυτό διαφάνειας λοιπόν εισάγουμε την διαφάνεια και έχουμε λοιπόν δύο καλές εκθέσεις και νομίζω πως ε, θα γίνουν και νόμος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάφ έχει ζητήσει το λόγο. Και μετά ο κύριος President... Ε, Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία έχετε γράψει εδώ πέρα. Σε γενικές γραμμές είμαστε σε καλό δρόμο και η διοργανική συμφωνία είναι βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν. Δύο ερωτήσεις έχω όμως όσον αφορά τους δικηγόρους και τους ιερείς. Ε, δεν είναι ακριβώς η ίδια ερώτηση αλλά γιατί και οι δικηγόροι και οι ιερείς καμιά φορά εργάζονται ως λομπίστες. Και καμιά φορά δίνουν ε, συμβουλές ε, στην περίπτωση δηλαδή των δικηγόρων και οι δε εκκλησίες είναι σε αυτόν τον ε, προνομιούχο διάλογο που αναφέρεται στη συνθήκη. Ξέρετε πως υπάρχει ένας επίσημος ε, διάλογος με τις εκκλησίες όπως ακριβώς ε, με τους εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων. Δεν είναι απλή λομπίστες. Έχουν λοιπόν δύο ρόλους και δύο ξεχωριστές λειτουργίες. Και νόμιζα, αν ναι, και δεν το έχω τώρα πρόχειρο, πως στην διοργανική συμφωνία υπάρχει διάκριση μεταξύ των ε, λειτουργιών αυτών ανθρώπων, των ρόλων τους. Και στο ψήφισμά μας, στην παράγραφο 6, β, ε, η διάκριση αυτή δεν γίνεται όσον αφορά τους ιερείς. Οι δε δικηγόροι δεν αναφέρονται και αυτό νομίζω είναι λάθος. Οπότε ήθελα κάποιες διευκρινήσεις εδώ πέρα. Όσον αφορά δε τον κανονισμό στην τροπολογία 5 Δεν καταλαβαίνω που το πάμε. Τι παράγραφο αυτή. Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα. Κάποιος, κάποιου ο οποίος έχει δελτίο μακροχρόνιο, μακροχρόνιο δελτίο εισόδου. δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της συμφωνίας. ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός αυτό. Η δημοκρατία χρειάζεται διαφάνεια και πρέπει να κάνουμε κάθε, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να μην δημιουργηθεί η εντύπωση πως γίνονται εδώ πέρα μυστικές συμφωνίες, διάφορες δουλειές ύποπτες και δεν μπορεί και, δε και ασκείται κάποια αθέμητη επιρροή στους βουλευτές. Οπότε το μητρό αυτό δεν είναι ικανή συνθήκη για τη διαφάνεια στην πολιτική η πρόσβαση στους βουλευτές, στους επιτρόπους, στην Κομισιόν είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να δείξουμε πως ε, υπάρχει διαφορετική πρόσβαση. Εμείς παλέψαμε για ένα τέτοιο μητρό διαφάνειας, οπότε θεωρούμε πως είναι μεγάλη επιτυχία, ακόμα και αν η τωρινή πρόταση βεβαίως δεν εκπληρώνει όλα όσα θέλαμε. όλα αυτά θα την υπερψηφίσουμε γιατί χαιρόμαστε γι' αυτό το μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω πως ε, δεν ρυθμίζονται εδώ πέρα όλα τα ζητήματα, πάρα πολλά παραμένουν ανοιχτά, δεν καλύπτεται το Συμβούλιο και θεωρούμε πως υπάρχει και η ίδια ανάγκη εδώ πέρα όπως ε, και για την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και το δεύτερο είναι πως ε, η καταγραφή αυτή δεν είναι υποχρεωτική στο Μητρό αυτό είναι έλλειψη και θεωρώ πως η έλλειψη αυτή δεν θα θεραπευτεί με το να λέμε ότι όποιος ε, δεν θα το κάνει δεν θα έχει μπάτζ ε, μακράς διαρκείας αυτό εύκολα γίνεται να βγάλει κανείς μπάτζ επίσης δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε συναντήσεις εκτός ε, του κτηρίου. Σε άλλα ε, οργανωτικά επίπεδα. Αυτά δεν μπορούμε να τα ρυθμίσουμε τυπικά όσον αφορά τη συμπεριφορά μας. Ε, και βεβαίως ο κάθε βουλευτής είναι και παραμένει... Πώς να πω υποχρεωμένος να ακολουθήσει μια ηθική που θα ξεδιαλύνει κάθε υποψία. Αλλά χαιρετίζουμε το αποτέλεσμα. Βεβαίως θα θέλαμε περισσότερα, αλλά έτσι είναι τα πράγματα στην πολιτική. Οπότε συμφωνούμε. Yeah, im Anschluss... Ναι. Γι' αυτό το οποίο είπε ο Άντριου Νταφ για το 6β εδώ πέρα αποκλείονται οι κοινωνικοί εταίροι, οι εκκλησίες και έχουμε δύο ομάδες που δεν θα τις λέγαμε ομάδες συμφερόντων αυτοί οι οποίοι έχουν δημόσια αξιώματα, αυτοί είναι οι συμβολεογράφοι, όπου αυτό θεωρείται δημόσιο αξίωμα, και οι δικαστές. Ε, δεν είναι δυνατόν νομίζω να χαρακτηρίσουμε λομπίστες στους δικαστές ε, όταν πρόκειται για την ε, δικαστική εξουσία δεν μπορώ, νομίζω αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε λομπίστες θα ήθελα λοιπόν να επανεξετάσετε πως μπορούν να εξαιρεθούν αυτές οι δύο ομάδες γιατί όταν μιλάμε για εκεί που έχουμε δημόσιο αξίωμα για μένα εξορισμού δεν μπορούμε να μιλάμε για λομπίστες ε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν μιλάμε λοιπόν για τη δικαστική εξουσία και συμβολεογράφους οι οποίοι είναι ε, οι οποίοι είναι λειτουργοί της δικαιοσύνης δεν νομίζω να μπορούμε να τους περιλάβουμε εδώ πέρα. Ε, thank you. This isn't so much a comment. Ευχαριστώ. αυτό δεν είναι τόσο σχόλιο, περισσότερο ερώτηση, διευκρίνηση που ίσως δεν ξέρω σας κάνει να, σας σκεφτείτε πως δεν το διάβασα πάρα πολύ καλά μια ματιά έριξα όπως κατάλαβα προσεγγίζεται το πρόβλημα του λόμπινγκ και από τις δύο πλευρές δηλαδή κοιτάτε τις οργανώσεις οι οποίες ε, αναμφισβήτητα είναι λόμπι με γνωστά συμφέροντα προκαταλήψεις και δεσμεύσεις και μετά εξετάζετε το πώς συμπεριφέρονται και έχετε κάποιες προδιαγραφές από την άλλη όμως εδώ θα έπρεπε να συμπεριλάβετε νομίζω πιστοποιημένους και τοπικούς βοηθούς που οπωσδήποτε θα επηρεάσουν την νομοθεσία. Και μετά θα έπρεπε να δείτε αυτοί μήπως έχουν κάποιες άλλες ε, επιρροές. Αυτό θα κάνετε. Αυτή την, ε, την ευκρίνηση έχω χωρίς να σημαίνει ότι ε, είμαι υπέρ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Εγώ ήθελα στη διάρκεια της συζήτησης και έγκρισης της υπόθεσης αυτού του κοινού Μητρώου να προβάλλουμε λίγο και την πολιτική σημασία πέρα από το θέμα της νομοθεσίας και του κανονισμού που έχει το θέμα αυτό. Βρισκόμαστε εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης η οποία σε πολλές χώρες ε, οδηγεί σε επιδύναμση της κοινωνικής αξίας των θεσμικών οργάνων και πιο συγκεκριμένα των κοινοβουλίων. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτή τη στιγμή Προσπαθούν να εισαγαγούν αυστηρότερους μηχανισμούς, μηχανισμούς διαφάνειας, συμβατότητας, απαγορεύσεις ε, στους βουλευτές τους σε εθνικό επίπεδο. Και επίσης, πολύ συχνά κατηγορείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι λαμβάνει μέτρα περιοριστικού χαρακτήρα, κάνει περικοπές ε, οι οποίες ε, υποχρεώνονται να κάνουν ε, πολλές ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κρίσης. Και έτσι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι ουσιαστικά στο στόχαστρο των παραπώνων και της ε, δυσαρέσκειας των Ευρωπαίων πολιτών Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι εμείς ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και θα πρέπει να το δούμε και από πλευράς ε, ηθικού αλλά και πολιτικού μηνύματος που πρέπει να περιλαμβάνει. Εγώ θεωρώ ότι η διαφάνεια είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την απαγόρευση. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες οι οποίες ε, ε, επισημαίνουν ότι όταν δημοσιοποιεί κάποιος αυτό που κάνει περιορίζει περισσότερο την απαγόρευση διότι υπάρχουν πάρα πολλοί που βρίσκουν μηχανισμούς για να παρακάμψουν τις απαγορεύσεις. Όταν εγώ ξεκίνησα να εργάζομαι ως δημόσιος υπάλληλο στην Ισπανία πριν από πάρα πολλά χρόνια, είχα και μαλλιά τότε, υπήρχε μια αγγλική έκφραση που έλεγε ότι όταν επιλέγεις δημόσιους λειτουργούς, το πιο σημαντικό είναι να είναι τίμοι. Διότι αν δεν είναι τίμη όσο περισσότερο γνωρίζουν, τόσο το χειρότερο. Που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι όλα στην επιφάνεια αυτά που γίνονται, διάφανα και να μην υπάρχει ένας επιπλέον κατάλογος απαγορεύσεων, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι όποιος παραβιάζει τους κανόνες της διαφάνειας, όπως ε, τόνισε ο Ματίας Γκρότε, θα έχει σαφείς και σημαντικές συνέπειες. Και τέλος, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη συμφωνία, αλλά είμαι πεπισμένος ότι αυτή τη στιγμή ε, θα προχωρήσει το κοινό μητρό μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πιεστεί και το Συμβούλιο με τον ένα με τον ένα άλλο τρόπο για να συμμετέχει και αυτό στη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Chair. Just a brief thought. Ευχαριστώ. Μία σύντομη σκέψη, Πρόεδρε. Εξάλλου, όταν συζητούσαμε την έκθεση του, το είχα πει αυτό. Λοιπόν, Πρώτον, το θέμα, το πρόβλημα με τη διαφάνεια είναι ότι είναι ασαφή τα σύνορα. Πότε δηλαδή γίνεται επικίνδυνη η εκπροσώπηση των ε, ε, ειδικών ομάδων, των εκπρόσωπων συμφερόντων. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν διάφοροι που ασκούν τέτοια δραστηριότητα. Οι διπλωμάτες επίσης ορισμένες φορές ασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες. Ε, οπότε πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε τη διάκριση. Δεν λέω ότι υπάρχει τίποτα επιλήψιμο στην διατύπωση που έχουμε επιλέξει, αλλά βάσει ε, των κανόνων διαφάνειας ε, που είναι ασαφής θα πρέπει να το προσέξουμε για να οριοθετήσουμε καλύτερα το, το κείμενο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι μεταξύ αυτών που επιδοκιμάζουν την πρόοδο που σημειώνεται. Βέβαια, ε, πιστεύω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά. Ε, ούτως ή άλλως, ε, θα επανέλθουμε στην εξέταση αυτού του κειμένου και θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Δεν θα ολοκληρωθούν σήμερα, αλλά πάντως θεωρώ ότι πρέπει να εξεταστεί το θέμα πριν τις επόμενες εκλογές, ευρωπαϊκές εκλογές. Καλό θα ήταν να γίνει μια αναθεώρηση πριν τις εκλογές, ώστε οι ψηφοφόροι να εμπλακούν ε, πλήρως ε, στις συζητήσεις για αυτό το θέμα. Κατά τη γνώμη μας ε, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τους πόρους που μπορούμε να αφιερώσουμε ε, στην μεταχείριση των εκπροσώπων συμφερόντων. Κατόπιν, ε, το Μητρό καταρτίζεται σε θελούσια βάση. Αλλά αναρωτιέμαι ποιες είναι οι κυρώσεις που προβλέπονται. Φαντάζομαι ότι η ίστατη κύρωση θα είναι να αποβληθεί κάποιος, να διαγραφεί από αυτό το Μητρό, το οποίο φαντάζει σοβαρό. Πάντως στα πλαίσια της αναθεώρησης ε, που προανέφερα καλό θα ήταν να εξετάσουμε και αυτό το θέμα της μη τήρησης των κανόνων. Παραδείγματο χάρη, όταν κάποιος ε, καταθέσει πλημελείς ε, πληροφορίες στο Μητρό δεν θα έπρεπε να διαγραφεί απαραίτητα από το Μητρό αλλά θα έπρεπε όλοι να ενημερωθούν ότι είναι εσφαλμένες οι πληροφορίες. Αυτά και τα υπόλοιπα κοινά, νομίζω κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα ε, διαλευκανθούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τις περισσότερες απόψεις που ακούστηκαν για το Μητρό της ε, Διαφάνειας και την Διοργανική Συμφωνία η οποία εντωμεταξύ επετεύχθη. Θεωρώ όμως πως δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που αντιλαμβάνονται πλήρως το πώς ε, θα είναι η επίδραση σε εθνικό επίπεδο και συγκεκριμένα στα νέα κράτη-μέλη. Για καιρό εμάς ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες. Μιλούσαν για καπιταλισμό, για τα λόμπι, σαν κάτι αρνητικό. Και εξακολουθούν να υπάρχουν ε, ακόμα παρανοήσεις ως προς αυτούς τους όρους. Γι' αυτό θα πρέπει νέα αυτή πρόταση να θεωρηθεί κάτι το το νέο και όχι οπωσδήποτε ως μια υπόθεση ρουτίνας. Χαίρομαι για το ότι θα έχουμε και στα νέα κρατημέλη αυτό το Μητρό και θα εργαστούμε στο πλαίσιο αυτού του Μητρώου. Είμαι πεπισμένος πως είναι αναγκαίο λοιπόν οι πολίτες μας να ξέρουν με λεπτομέρειες τα του Μητρώου αυτού και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να αναφέρω και τα ΜΜΕ. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης γιατί και αυτοί ενημερώνουν την κοινωνία, την κοινή γνώμη και καμιά φορά διαδίδουν σωστές πληροφορίες, άλλες φορές λανθασμένες πληροφορίες. Και θα πρέπει και αυτούς ως ένα βαθμό να τους θεωρήσουμε λομπίστες. Οπότε προσοχή και στα μήμια παρακαλώ. Καλώς. Μπορείτε να εκφράσετε τις επιφυλάξεις σας μέσω τροπολογιών. Προτείνω να ψηφίσουμε αυτές τις δύο εκθέσεις στις 19 Απριλίου και θα ήθελα να θέσω την προθεσμία για την παρουσίαση τροπολογιών στις 24 Μαρτίου τα μεσάνυχτα, ώστε να έχετε χρόνο να εκφράσετε και επισήμω ε, τα αιτήματά σας για προσθήκες ή διορθώσεις. Θα ήθελα τώρα να κάνω μια απόπειρα να απαντήσω σε κάποιες από τις παρεμβάσεις σας. Καταρχάς, να σας πω ότι ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, κύριε Χέφνερ, πώς είναι δυνατόν να ε, θέλουμε να έχουμε ένα υποχρεωτικό μητρό. Τι σημαίνει υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό θα σημαίνει ότι όλες ε, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και όχι μόνο βελγικές όλες οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να εγγραφούν σε ένα μητρό ακόμα και αν δεν το χρησιμοποιήσουν ποτέ και δεν έρθει κανείς ποτέ εδώ. Ε, δεν μπορούμε να τη θέσουμε έτσι την υποχρέωση. Η υποχρέωση σημαίνει ότι οποιοδήποτε θέλει να έχει σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προασπίσει τα συμφέροντά του θα πρέπει και υπ' αυτή την έννοια είναι υποχρεωτικό, αλλά από τεχνική άποψη βάση του Ιταλικού δικαίου και εν γέννη δεν μιλάμε για υποχρέωση αλλά για χρέος. Έχω καθήκον να σέβομαι κάποιους ε, κανόνες αν θέλω να απολαμβάνω κάποιων εκτιμάτων. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα περιλαμβάνονται σε συμφωνία εγώ για λόγου συντομία δεν σα τα διάβασα, αλλά μπορείτε να τα βρείτε στη συμφωνία. Υπάρχει και ένα κώδικα διοντολογία ο οποίο ισχύει. Εννέα σημεία τα οποία ισχύουν για όλου όσου θέλουν να εγγραφούν στο Μητρό. Επομένω δεν πρόκειται ε, διαφάνεια κατόνομα, πρόκειται για μία δέσμευση να σεβόμαστε τη διαφάνεια. Επομένω, υπάρχουν και κάποιε συγκεκριμένε υποχρεώσει. Αυτό όσον αφορά το θέμα του υποχρεωτικού ημί. Το Μητρό είναι χωρισμένο σε διάφορα τμήματα, μπορείτε να τα δείτε στη συμφωνία. Έχουμε έξι διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες ουσιαστικά δεν κάνουν τόσο διαφοροποίηση ως προς τη μεταχείριση, διότι όλοι είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τον κώδικα διοντολογίας. Κάνω μια διαφοροποίηση μεταξύ της επιχείρησης που προσπαθεί να έχει κάποια οικονομικά ωφέλη και του πολιτιστικού ιδρύματος που θέλει να συνεισφέρει στην Ευρωπα... στον ευρωπαϊκό πολιτισμό προσφέροντας ιδέες, προτάσεις και παρακολουθώντας λίγο πιο επισταμένα τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα θεσμικά όργανα εν γέννη για να βοηθήσει στο όλο ε, οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό έχουμε και έξι διαφορετικές κατηγορίες. Έχουμε τους εμπορικού, για παράδειγμα, φορείς που είναι σε διαφορετική κατηγορία από τους δικηγόρους. Οι νομικοί φορείς ούτως ή άλλως είναι τελείως διαφορετικοί από τους πολιτιστικούς φορείς, διότι ε, τα δικηγορικά γραφεία μπορεί να είναι και εκπρόσωποι πολύ ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Επομένως, ε, υπάρχει μια διαφοροποίηση. Όσον αφορά τώρα την παρουσία της Εκκλησίας ε, στο Μητρό, ε, τους έχουμε στην πέμπτη κατηγορία, βάσει του άρθρου 17, δεν κάνω λάθος, ε, της συνθήκης για την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι όμως η Εκκλησία αυτή καθεαυτή. Λέει στο κείμενο ότι έχουμε νομικά πρόσωπα γραφεία και δίκτυα τα οποία καθορίζονται μέσω της εκπροσώπησης. Επομένως, ο απλός, ε, ε, ο που θα έρθει εδώ υπόκειται στους συνήθεις κανόνες που ισχύουν για όλους. Και επομένως απαντώ και στο ποιο ε, μπορεί να έχει άδεια εισόδου και σε ποιον μπορούμε να δώσουμε δελτίο ελευθέρας εισόδου για άνω του ενός έτους αν δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό ε, αυτό το λέει η τροπολογία 3 στην παράγραφο 9 που λέμε ότι ο, το δελτίο δευτέρα εισόδου μπορεί να εκδοθεί για όσους θέλουν να έχουν πρόσβαση συχνά στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας για το Μητρό. Πιο συγκεκριμένα γίνεται διευκρίνηση για τους ε, τοπικούς βοηθούς των Ευρωβουλευτών. Παραδείγματο χάρη, εγώ όταν μπορώ ζητώ από τη γυναίκα μου να με συνοδεύει και έχει ένα δελτίο εισόδου που τη επιτρέπει να μπει και ξέρουμε ότι είναι συγγενή. Αυτό είναι μία περίπτωση. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε διάκριση λοιπόν μεταξύ των διαφόρων περιπτώσεων. Να απαντήσω και σε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Το Συμβούλιο, αυτό είναι σημαντικό, αλλά ευτυχώς αυτό είναι γραμμένο και στην ίδια τη συμφωνία. Σημείο 28, το οποίο προκύπτει από τη συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών καλούνται να προσχωρήσουν στη, στο Μητρό. Υπάρχει λοιπόν επίσημη πρόσκληση προς το Συμβούλιο και ελπίζουμε σύντομα να τη δεχθούν την ε, πρόσκληση. Οι κυρώσεις τώρα. Ε, προβλέπονται κυρώσει. Είναι λογικό. Αν δεν σέβεται κάποιο τον κώδικα δεοντολογία και τι υποχρεώσει που απορρέουν από αυτό, υπάρχουν και κυρώσει οι οποίε είναι διαβαθμισμένε σε τέσσερι διαφορετικέ κατηγορίε. Υπάρχει κύρωση σε περίπτωση που κάποιο ε, κάνει ε, εκούσια ε, παρατυπία. Υπάρχει επίσης και η εσκεμμένη παρατυπία που, υπάρχει, ε, που έχει και συγκεκριμένη κύρωση υπάρχει και κατά παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας και τέλος υπάρχει και σοβαρή παρατυπία και παραβίαση του, κανόνα, του κώδικα δεοντολογίας και αυτό φυσικά ε, έχει και διαφορετικές διαβαθμίσεις της κυρώσεις από μία απλή ε, κοινοποίηση και παρατήρηση μέχρι ε, προσωρινή απαγόρευση πρόσβασης μέχρι και μόνιμη απαγόρευση πρόσβασης. Υπάρχουν λοιπόν τα κυρώσεις. Νομίζω ότι λίγο πολύ απάντησα σε όλες τις ενστάσεις σας. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να διαβάσετε τα έγγραφα και κυρίω την ε, συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, η οποία είναι πολύ πιο διεξοδική, η οποία θα σα επιτρέψει να παρουσιάσετε και τροπολογίε εντό ε, τη 24η Απριλίου τα μεσάνυχτα. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις μπορούμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν με το σημείο αυτό και να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. στο σημείο υπαριθμών 6 έχουμε την έκθεση DAF, την οποία έχουμε αναβάλει για αύριο. Επομένως, να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γιαννάκου, διότι το σημείο 7, η εφαρμογή του κανονισμού 2004-2003 για το καθεστώ και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η η κυρία Γιαννάκου. Θα θυμάστε ότι έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό και στις 26 Ιανουαρίου έγινε και σχετική ακρόαση, πολύ σημαντική, το σχέδιο έκθεσης παρουσιάστηκε από την εισηγήτριά μα στι 17 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ε, συνεδρίασης της Επιτροπής μας. Παρουσιάστηκαν 99 τροπολογίες. Δυστυχώς έχουμε στη διάθεσή μα τις τροπολογίες μόνο στην αγγλική γλώσσα. Θα ξεκινήσει η συζήτηση τώρα και θα δούμε αν από τη σημερινή συζήτηση θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε αύριο το πρωί στην ψηφοφορία όπως ε, επιθυμεί η εισηγήτρια. Παρακαλώ κυρία Γιαννάκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πράγματι η έκθεση αυτή είναι η επόμενη μετά την έκθεση που είχε γίνει το 2007 αφού τροποποιήθηκε ο κανονισμός το 2006 για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων που χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκά κεφάλαια κατά βάση ε, από ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η πρότασή μου ώστε τα κόμματα να αποκτήσουν ένα πραγματικό πολιτικό και νομικό καθεστώς διότι αυτή τη στιγμή τα κόμματα είναι ένα είδος διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης ε, πρώτον αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που επιτάσσει η συνθήκη της Λισαβόνας η οποία ομιλεί για το δημοκρατικό ρόλο των κομμάτων και τη σημασία τους μέσα στο χώρο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας ε, και δεύτερον διότι στην ουσία δεν μπορούν να υπάρξουν συνομιλητές οποιοδήποτε με το πολιτικό βάρος που χρειάζεται. Ο Γενικός Γραμματέας έχει πραγματοποιήσει, έχει συγγράψει μια έκθεση η οποία βασίζεται βέβαια στην χρηματοδότηση και τα αποτελέσματά της μέσα στα οποία είναι και τα συμπεράσματα του ελεγκτικού συνεδρίου. Επ' αυτής επίσης υπάρχει ένα σημείωμα του Μπυρό, το οποίο εξήτασε το θέμα. Και η έκθεση του 2007 ε, τόνιζε την ε, ε, υποχρέωση να έχουμε ένα πολιτικό, νομικό και φορολογικό καθεστώς για τα κόμματα. Και βεβαίως κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε κύριε Πρόεδρε στην Ακρόαση όπου όπως θυμάστε είχαμε καλέσει όλους τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων καθηγητές πανεπιστημίου το ελεγκτικό συνέδριο και τη διεθνή διαφάνεια. Ε, στη συζήτηση αυτή όλοι ε, ετώνησαν ότι δεν πρέπει να είναι μόνο μέλη των κομμάτων, των ευρωπαϊκών κομμάτων, εθνικά κόμματα ή περιφερειακά κόμματα, αλλά θα μπορούσαν και πρόσωπα, άτομα να γίνουν μέλη των κομμάτων αυτών και αυτό βεβαίως δεν μπορεί κανείς, όχι μόνο δεν μπορεί κανείς να το εμποδίσει, <clears throat> αλλά θα πρέπει να το ευνοήσει. Σημειώνω ότι μέλη των κομμάτων μπορούν να είναι τουλάχιστον και πρέπει να είναι σε 7 χώρες, ε, είτε μέλη κομμάτων που είναι εθνικά, και επομένως έχουν εκπροσώπηση στην Εθνική Βουλή, είτε μέλη κομμάτων που είναι περιφερειακά αλλά οι περιφερειακώς εκλεγμένοι θα πρέπει να έχουν νομοθετικές αρμοδιότητες. Σημειώνω ότι υπάρχουν χώρες όπως η Ισπανία ή η Γερμανία όπου ε, υπάρχουν περιφερειακά κοινοβούλια με νομοθετικές αρμοδιότητες. Στη δική μου χώρα υπάρχουν περιφερειακές αρχές χωρίς νομοθετικές αρμοδιότητες. Ε, επομένως ε, αυτό είναι μια σημαντική βάση. Απ' την άλλη πλευρά, στο θέμα της χρηματοδότησης, ε, θα πρέπει και μένουμε σε αυτό που ορίζει ο κανονισμός να υπάρχει τουλάχιστον ένα κόμμα, ένα μέλος εκλεγμένο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλοί εκ των συναδέλφων θέλησαν να διαχωρίσουν ε, το ποιο είναι Ευρωπαϊκό Κόμμα και αν χρηματοδοτείται. Και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό, δηλαδή θα μπορούσε κανείς να δώσει ταυτότητα ενός Ευρωπαϊκού κόμματος σε ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται πριν από τις ευρωεκλογέ, δημιουργείται για πρώτη φορά, αλλά δεν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί αν δεν εκλέξει τουλάχιστον ένα μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο ίδιο πλαίσιο κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν διάφορες τροπολογίες και προτάσεις για τη χρηματοδότηση. Βεβαίως η χρηματοδότηση μέχρι τώρα ήταν από πρόσωπα μπορούσαν να πάρουν τα κόμματα αυτά μέχρι 12.000 ευρώ. Άπαξ. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να διπλασιαστεί, να γίνει 25 υπό τις συνθήκες που βρισκόμαστε, 25 και όχι παραπάνω. Υπάρχουν επίσης προτάσεις από συναδέλφους ε, οι οποίες θεωρούν ότι επειδή τα ευρωπαϊκά κόμματα θα γράψουν και μέλη ε, θα πρέπει τα περισσότερα χρήματα να τα προσπορίζονται από τα μέλη τους. Αυτό κύριε Πρόεδρε δεν μπορώ να το δεχθώ και δεν είναι δυνατόν για τον πολύ απλό λόγο αυτό θα μπορούσε να είναι δυνατόν 10 χρόνια μετά παραδείγματο χάρη αν και όταν τα κόμματα αυτά αποκτήσουν και μέλη άτομα αλλά δεν είναι δυνατόν τα, ευρωπαϊκά κόμματα να συντηρηθούν παραδείγματο χάρη επειδή λίγοι άνθρωποι θα πληρώνουν από 20 ευρώ το χρόνο ε, ως ε, συμβολή στα ευρωπαϊκά κόμματα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ε, και όχι παράλογοι στο θέμα αυτό. Μη φύγουμε δηλαδή από μία γραμμή που θα βοηθήσει τα κόμματα να αποκτήσουν πραγματικά νομική και πολιτική προσωπικότητα και επομένως να συμμετέχουν και στις ευρωπαϊκές καμπάνιες και να έχουν ένα πραγματικό στάτους που μπορεί να τους κάνει σοβαρούς συνομιλητές. Σας θυμίζω ότι τα εθνικά κόμματα έχουν συγκεκριμένο νομικό στάτους ως κόμματα στα κράτη-μέλη. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ότι τα ευρωπαϊκά κόμματα μπορεί να είναι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Όσον αφορά στη διαχείριση κύριε Πρόεδρε, ε, δεν έχουν διαπιστωθεί ανομαλίες και προβλήματα. Λαμβάνουμε υπόψη μας βέβαια στην έκθεση και τις παρατηρήσεις που έκαναν και από το ελεγκτικό συνέδριο αλλά και από τη διεθνή διαφάνεια. Διότι ζούμε σε μια εποχή όπου η διαφάνεια έχει τεράστια σημασία. Τα μίντια και οι πληροφορίες που φτάνουν στους πολίτες και στους λαούς πολλές φορές δημιουργούν και διαστρεβλωμένη εικόνα και καλό είναι να φροντίσουμε να είμαστε άψογοι ε, στα θέματα που αφορούν στη δημοσιότητα και στη διαφάνεια σε σχέση με τα κόμματα. Ζητάμε τελικά κύριε Πρόεδρε να ε, υπάρξει μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αποκτήσουν τα ευρωπαϊκά κόμματα ταυτότητα και να μπορούν παραδείγματο χάρη στις συζητήσεις που κάνουμε το βελγικό κράτος γιατί είναι εγκατεστημένα εδώ στο Βέλγιο να έχουν νομική προσωπικότητα, να έχουν φερεγγιότητα αφού μάλιστα χρηματοδοτούνται από ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χρηματοδοτούνται δηλαδή με ευρωπαϊκά κεφάλαια. Στην πραγματικότητα, επί της ουσίας, έχουμε αναγνωρίσει το ρόλο των κομμάτων αυτών, πολλά από τα οποία έχουν δύο δεκαετιών τα έχουμε αναγνωρίσει διότι τα χρηματοδοτούμε. Έχουμε αναγνωρίσει επίσης τα ιδρύματα που προέρχονται από τα κόμματα ε, όπου εδώ άλλες ε, ε, τροπολογίες τα θέλουν affiliated, άλλες αλλιώς. Εγώ έχω σημειώσει στις τροπολογίες, τις συμβιβαστικές που έχουν γίνει ότι είναι κόμματα όπως ακριβώς τα περιγράφει ο κανονισμός και ο κανονισμός τα περιγράφει affiliated είτε their foundations είτε ε, with ε, their affiliated foundations ε, είναι το ίδιο πράγμα. Τα ιδρύματα κύριε Πρόεδρε προσφέρουν πολύ καλές υπηρεσίες όχι μόνο στα κόμματα αλλά και γενικότερα στις πολιτικές ομάδες που είναι μέσα στο κοινοβούλιο, στα πολιτικά groups δηλαδή αφού προβαίνουν σε διάφορες εκδηλώσεις προς διάφορες κατευθύνσεις, κυρίως όσο αφορά την εφαρμογή των κανόνων της δημοκρατίας, τη διαφάνεια, την απελευθέρωση διαφόρων πολιτικών, τις συζητήσεις γύρω από ιδεολογικά και άλλα θέματα, μέσω της οποίας και η συμμετοχή εκπροσώπων τρίτων χωρών και ειδικά χωρών όπου δεν υπάρχει ευρωπαϊκού τύπου δημοκρατία συμμετέχουν. Άλλωστε η έκρηξη στο νότο της Μεσογειακής Ένωσης εναντίον των αυταρχικών καθεστώτων κύριε Πρόεδρε μας δίνει όλα τη δυνατότητα να πούμε με σιγουριά ότι τα ιδρύματα αυτά θα προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερες υπηρεσίε και ταυτόχρονα βέβαια και προς την πλευρά της ανατολικής συνεργασίας και προς χώρες που είναι ε, υποψήφια μέλη. Ε, δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο κύριε Πρόεδρε. Εγώ ζητώ να υπερψηφιστεί η έκθεση αυτή. Ξέρω ότι υπάρχουν ενστάσεις για το σημείο στο οποίο έχω ζητήσει και για το staff των κομμάτων να υπάρξει ένα νομικό και φορολογικό καθεστώς γιατί υπάρχουν συνάδελφοι από διάφορες πολιτικές ομάδες που έχουν υποβάλει τροπολογία αυτό να διαγραφεί. Φυσικά αυτό είναι μέσα στις ελευθερίες και τα δικαιώματα όλων μας. Εμένα αυτή είναι η πρότασή μου και νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι θα μπορέσουμε αύριο να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή και να επιδιώξουμε να επιταχύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαδικασίες για να έρθει μια πρόταση συγκεκριμένη για το στάτους των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνθήκη της Λισαβόνας πλέον ε, έχει 1,5 χρόνο που ε, λειτουργεί και επομένως θα πρέπει να ανταποκριθούμε στα κελέσματα της συνθήκης και στο γεγονός ότι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νομική προσωπικότητα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν τα πολιτικά κόμματα που έχουν νομική προσωπικότητα στα κράτη-μέλη ε, να είναι χωρίς νομική προσωπικότητα σε επίπεδο ένωσης. Αυτό απαιτεί νομίζω η δημοκρατική τάξη και η σημερινή πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία κύριε Πρόεδρε και σας προσωπικά ε, για τη βοήθεια και για την πραγματοποίηση αυτής της ε, ακρόασης η οποία νομίζω προσέθεσε σημαντικά στις σκέψεις μας προκειμένου να γίνει αυτή η έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ κυρία Γιαννάκου, όχι μόνο για την παρέμβασή σας, αλλά και για την τεράστια δουλειά που κάνατε. Ο κύριος Γκερέρο έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Γιαννάκου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση που κάνατε σήμερα, αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος μας, σας ευχαριστώ πολύ και για το τεράστιο έργο που κάνατε στη διάρκεια ε, της ε, επεξεργασίας αυτής της έκθεσης. Νομίζω ότι στην Επιτροπή μας ε, συμφωνούμε ότι οι πολιτικές ομάδες, τα πολιτικά κόμματα είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την ε, αντιπροσωπευτική δημοκρατία και η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι το επίκεντρο των θεσμικών μας οργάνων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορούμε να την εμπλουτίσουμε και να τη συμπληρώσουμε και έτσι θα γίνει με την ε, νομοθετική πρωτοβουλία που εγκρίναμε πριν από κάποιους μήνες χάρη στις ε, προσπάθειες της κυρίας ε, Σίτα Φωνμάη και του κυρίου Λαμασούρ. Η γενική θεωρία για τα πολιτικά κόμματα λέει ότι είχαμε τέσσερις μεγάλες ε, σημαντικές στιγμές στην ιστορία από τις ε, επαναστάσεις των εργατών μέχρι το ε, καθεστώς αυτών των πολιτικών κομμάτων. Το πρώτο στάδιο ήταν η απόρριψη των κομμάτων, το δεύτερο στάδιο ήταν η άγνοια για τα πολιτικά κόμματα, το τρίτο στάδιο ήταν η νομιμοποίηση των πολιτικών κομμάτων και το τελευταίο στάδιο ήταν ε, το γεγονό ότι πλέον είναι θεσμικά, ε, θεσμικό δικαίωμα τα πολιτικό κόμματα και όλοι στις χώρες μας ε, ξέρουμε ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν διεξάδει ένα σημαντικό ρόλο στην σχηματισμό της κοινή γνώμης και την συμμετοχή στα κοινά των πολιτών. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει δώσει πλέον καθεστώς στα πολιτικά κόμματα και Προσπαθούμε τώρα να το συμπληρώσουμε και να το εμπλουτίσουμε αυτό το καθεστώς, δίνοντας ένα νομικό καθεστώς στα πολιτικά κόμματα και ξεπερνάμε πλέον το στάδιο και δεν θεωρούμε τα πολιτικά κόμματα ως κάτι το οποίο είναι ξένο προς την ε, θεσμική διαδικασία και ε, πλέον λαμβάνουν ένα νομικό καθεστώς. Έχουμε 99 τροπολογίες για την έκθεσή σα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται για μία έκθεση την οποία αμφισβητεί η πλειοψηφία της Επιτροπής μας. Το αντίθετο. Θεωρώ ότι υπάρχει συνένεση σε πολύ μεγάλο βαθμό μεταξύ των μελών της Επιτροπής. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη συνένεση, διότι έγινε μια προπαρασκευαστική εργασία με τα μέλη της Επιτροπής, με τις πολιτικές ομάδες ε, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με εκπροσώπους που ήρθαν εδώ. Επομένως αυτές οι 99 τροπολογίες δεν δικαιολογούν το υψηλό επίπεδο συνένεσης που έχουμε αυτή τη στιγμή για την έκθεσή σας. Η ομάδα μου παρουσίασε τροπολογίες μέσω εμού, μέσω του κ. Ματίας Ρότα, της κυρίας Σίτα ε, τον κύριο Γιάννεφ, ε, έχουμε παρουσιάσει μια σειρά από τροπολογίες τις οποίες θα προσπαθήσω να εξηγήσω. Να σταθώ λίγο στην ουσία. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες ε, που έχουν σχέση με την αιτιολογική σκέψη ΑΑ και το άρθρο 10 και αναφέρονται στη διαγραφή, στην αναφορά στην έκθεση στο φορολογικό καθεστώς για το προσωπικό των ε, πολιτικών κομμάτων. Να σας πω ότι δεν είναι αντίρρηση επί της αρχής, απλώς ε, σκεφτόμαστε λίγο την πολιτική συγκυρία που βιώνουμε και τη δυσκολία που θα είχαν ε, πολλοί να εξηγήσουν αυτή τη το φορολογικό τους καθεστώς για τους υπαλλήλους, για τους εργαζόμενους, για τους ανθρώπους που αποσχολούνται από τα πολιτικά κόμματα στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε τη ρύθμιση αυτού του θέματος σε κάποια μελλοντική στιγμή, αλλά θα προτιμούσαμε να μην γίνει αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε κατά, απλώς θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό στην έκθεση ε, τη συγκεκριμένη, διότι θα ήταν πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στην κοινή γνώμη ε, το θέμα από πολιτική σκοπιάς. Υπάρχει μια άλλη τροπολογία η οποία αφορά τη διαφοροποίηση μεταξύ των προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος και των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων για τη χρηματοδότησή του η ομάδα μας θεωρεί ότι τα πολιτικά κόμματα μπορούν να συσταθούν με διαφορετικές προϋποθέσεις, ε, με διαφορετικό τρόπο, ε, ανάλογα με τις προτιμήσεις αυτών που θα αποτελούν αυτό το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα και θα πρέπει να τηρούνται και κάποιες προϋποθέσεις. Πολλές εξ αυτών περιλαμβάνονται στην έκθεση. Να υπάρχει εσωτερική δημοκρατική συμπεριφορά, να υπάρχουν κάποιες διαδικασίες συγγραφής και ούτω καθεξής. Αλλά δεν μπορούμε να απαιτούμε από ένα πολιτικό κόμμα το οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί στον ευρωπαϊκό χώρο, ότι για να είναι πολιτικό κόμμα θα πρέπει προηγουμένως να έχει εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, θα μπορούσε να μην έχει παρουσιαστεί κάποιο ως υποψήφιο στι ε, προηγούμενες ευρωεκλογέ. Η δημιουργία λοιπόν ενός πολιτικού κόμματος και η χρηματοδότηση είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ε, για τη μία περίπτωση δεν απαιτείται κανένας εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ για την εκπροσώπηση, για τη χρηματοδότηση απαιτείται τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, η η αιτιολογία είναι ότι δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε όλα τα πολιτικά κόμματα που σχηματίζονται, αλλά θα πρέπει μέσω μιας εκλογικής διαδικασίας να μας αποδείξουν ότι υπάρχει μια κάποια υποστήριξη για το συγκεκριμένο κόμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια άλλη τροπολογία τώρα αναφέρεται στο γεγονός ότι εμείς ε, θεωρούμε ότι πολλά σημεία της έκθεσής σας, πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 12, 14, 15 και 17, τα οποία αναφέρονται σε εκλογικές μεταρρυθμίσεις στον εκλογικό νόμο και στη διαδικασία εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε αυτή την έκθεση και σε αυτόν τον κανονισμό. Εδώ συζητάμε το καθεστώς των πολιτικών κομμάτων και τη χρηματοδότηση των ε, πολιτικών κομμάτων και όχι το κατά πόσον το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να είναι με τη μία ή με την άλλη μορφή, θα πρέπει να ε, τροποποιηθεί ε, το υφιστάμενο σύστημα και ούτω καθεξής. Το θέμα αυτό ούτως ή άλλως αναφέρεται στην έκθεση του κυρίου Νταφ και θεωρούμε ότι εκεί είναι ο καταλληλότερος χώρος για να ασχοληθούμε με πιθανές τροποποίησεις του εκλογικού συστήματος. Και όχι ο νόμος για το καθεστώς των πολιτικών κομμάτων, διότι στην ε, πλειονότητα των χωρών μας υπάρχουν πολιτικά κόμματα και υπάρχει και εκλογικός νόμος, ο οποίος δεν αφορά τον κανονισμό των πολιτικών κομμάτων. Επίσης, εμείς παρουσιάζουμε μια τροπολογία με την οποία λέμε ότι το καθεστώς των πολιτικών κομμάτων θα προσαρμοστεί στις μεταρρυθμίσεις που θα, μπορέσουν, θα μπορούσαν ίσως να παρουσιαστούν στο εκλογικό σύστημα. Δηλαδή, ε, εάν υπάρξουν αλλαγέ στο εκλογικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαν να γίνουν και αλλαγές για το καθεστώς των πολιτικών κομμάτων. Υπάρχει μια τροπολογία που αναφέρεται στο όριο των δωρεών Εμείς λέμε τα 25.000 ευρώ να είναι αναέτος και αναδορητή, αναχωρηγό. Και φυσικά θα πρέπει να υπόκειται και στην ισχύουσα νομοθεσία για τη διαφάνεια. Πρώτο τελευταίο σημείο. Λέμε ότι δεν είναι απαραίτητο τα πολιτικά κόμματα να συγχρηματοδοτούν στον ίδιο βαθμό με τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δηλαδή, στην Εθνική Νομοθεσία για τη Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων δεν απαιτείται συγχρηματοδότηση των ε, εθνικών κομμάτων για να λάβουν χρηματοδότηση ε, για τις εκλογές ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο. Εδώ παρουσιάζονται δύο τροπολογίες από τη σοσιαλιστική ομάδα η μία ζητά να μην υπάρχει το θέμα της χρηματοδότησης και η άλλη λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει μία μείωση κατά 10% σε σχέση με το 5% ε, που έχει έκθεση. Τέλος, ή μάλλον σχεδόν τελευταία παρατήρηση, γιατί έχω και μια τροπολογία τελευταία που θα ήθελα να θίξω. Εμείς θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε θέση για ε, το καθοστός ε, της εσωτερικής ε, κατάστασης affiliate σε ένα πολιτικό κόμμα. Το να λέμε ότι θα πρέπει κάποιος να ανήκει σε ένα εθνικό πολιτικό κόμμα για να μπορεί να ανήκει και στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, αλλά υπάρχουν και άλλες θέσεις που λένε ότι μπορεί κάποιος να ανήκει σε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα χωρίς να πρέπει να ανήκει στο αντίστοιχο εθνικό κόμμα. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να το αφήσουμε αυτό στην διακριτική ευχέρεια κάθε ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα θα καθορίζει πώς μπορεί κάποιο να ανήκει στο κόμμα. Αν θέλει κάποιο υποχρεωτικά να ανήκει σε εθνικό πολιτικό κόμμα προηγουμένω, μπορεί να το δεχτεί έτσι. Αν θέλει να μπορεί κάποιο να ανήκει στο κόμμα το ευρωπαϊκό χωρίς να είναι υποχρεωμένο να ανήκει στο αντίστοιχο εθνικό, Α το καθορίσει έτσι. Δεν θα καθορίζουμε εμεί πώ θα είναι ε, το εσωτερικό σύστημα εγγραφή στο κόμμα. Τέλο υπάρχει μια τροπολογία της κυρίας ε, Γκουρμάη, την οποία θα ήθελα να τη συνδέσω με την τελευταία, το τελευταίο τμήμα της παρέμβασης τη κυρίας Γιαννάκου, που αναφέρεται στη σημασία των ιδρυμάτων των ε, ε, ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και τη σημασία τους σε στιγμές στις οποίες η προάσπιση της δημοκρατίας, η διαβίβαση των γνώσεών μας, οι διαδικασίες μετάβασης είναι πολύ σημαντικές και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ε, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και τα ιδρύματά τους, συγγνώμη, διορθώνει ο μιλητής, ε, μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, να σας περιγράψω λίγο την ισπανική μου εμπειρία που είμαι βέβαιος ότι είναι σχεδόν η ελληνική εμπειρία της κυρίας Γιαννάκου και η πορτογαλική εμπειρία του κυρίου Ρενκέλ που είναι όλοι στην ίδια σειρά. Όλοι συμμετέχουμε στη διαδικασία πολιτικής μετάβασης και ξέρουμε τι υποστήριξη έχουμε λάβει από ιδρύματα, από ε, ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, ε, τα οποία είναι ιδεολογικά προσκύμενα στα δικά μας. Σε εσωτερικό επίπεδο αυτό θα πρέπει να είναι και ο κανόνας συμπεριφοράς ε, για περιοχές του κόσμου που βρίσκονται σε αυτές τις μεταβατικές διαδικασίες. Γνωρίζω ότι η κυρία Γιαννάκου παρουσίασε σήμερα το απόγευμα κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες Είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε τις περισσότερες εξ αυτών των συμβαστικών τροπολογιών και όπως και να έχει, όπως σας είπα, νομίζω ότι υπάρχει γενικότερη συνένεση για την έκθεσή σας και αύριο θα ψηφίσουμε και σε κάποιες περιπτώσεις θα σας υπερψηφίσουμε, σε κάποιες περιπτώσεις θα σας καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Um, um, Πρόεδρε, ναι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη σκληρή δουλειά της, γιατί είναι όντως σκληρή αυτή η δουλειά. Να σκάβει κάποιος κάτω από τις δομές των πολιτικών κομμάτων στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. βλέπει κάποιος σοβαρές διαφορές ως προς το καθεστώς, τις διαδικασίες, τη χρηματοδότηση, την κουλτούρα κάθε κόμματος και το καθεξής. το να ε, δημιουργήσει κάποιος ε, μια ευρωπαϊκή διατύπωση για ένα διεθνικό κόμμα δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Και θεωρώ ότι η κυρία Γιαννάκου τα καταφέρνει μία χαρά. Κυρίως με τις συμβαστικές της τροπολογίες που θα υποστηρίξω με μία μόνο εξαίρεση. Δύο σχόλια θα ήθελα να κάνω. Πρώτον, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε σύντομα να καταθέσει μία επίσημη νομοπαρασκευαστική πρόταση. Για την παράγραφο 18, την τωρινή παράγραφο 18, λέμε ότι καλείται η παρούσα επιτροπή να συντάξει μια επιπρόσθετη έκθεση που θα συμπεριλαμβάνει και νομοθετική πρόταση και η οποία κατόπιν θα υποβληθεί στην Επιτροπή. Ε, νομίζω ότι παρά είναι μακρά η διαδικασία που προβλέπετε και δεν χρειάζεται να είναι και τόσο βασανισμένη. Ας ζητήσουμε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει ένα σχέδιο καταστατικού δυνάμει και το άρθρο 225 της ε, συνθήκης. Προσπάθησα να το εκφράσω αυτό στην τροπολογία μου υπαριθμών 76. Εκεί περιγράφεται η ανάγκη ε, εκπόνησης νέας έκθεσης από την Επιτροπή Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει επαρκώς αυτό το θέμα ήδη. Το δεύτερο σημείο τώρα, και αυτό αναφέρεται στην συμβαστική G για την παράγραφο 31, δεν μπορώ να την υποστηρίξω αυτή την συμβαστική τροπολογία, μεταξύ άλλων διότι απευθύνεται έκκληση προς τις πολιτικές ομάδες να ε, δρομολογήσουν έναν προβληματισμό για το θέμα ε, του μέλους, ε, της ιδιότητας του άμεσου μέλους. Νομίζω ότι κανονικά εδώ και 20 χρόνια συζητείται αυτό το θέμα από τα, τις πολιτικές ομάδες και κανονικά θα έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει τη σκέψη τους. Αυτός είναι ο στόχο της τροπολογίας μου ε, παριθμών 97. Δηλαδή, ε, ζητάμε περαιτέρω εργασίες για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ε, ώστε να υπάρχει άμεση ιδιότητα άμεσου μέλους. Με έκφραση των προτιμήσεών τους βέβαια, όπως μας είπε και ο κύριος Γκερέρο δεν εξυπακούεται ότι σε όλες τις πολιτικές οικογένειες έχουμε όλοι πανομοιότυπη προσέγγιση για αυτό το θέμα. Αλλά θεωρούμε ότι έχει θεμελιώδη σημασία αυτό το ζήτημα. Για να αξιώσει κάποιος αυτό το καθεστώς του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος, ε, θα διευκόλυνε κάποιος την προσχώρηση νέων μελών, άλλων πολιτών. Άρα, στο καταστατικό του κόμματος θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικέ διαδικασίες, ούτως ώστε η... να υπάρχει ειδικό τμήμα για τους πολίτες που είναι μέλη του κόμματος, ούτως ώστε να μπορούν να μετάσχουν στις όλες τις διαδικασίες και συγκεκριμένα στη διαδικασία λήψη αποφάσεων των ε, κομμάτων. Θα ήθελα λοιπόν με μεγαλύτερη πυγμή να πιέσω προς την κατεύθυνση προς την οποία ούτως άλλως κατευθύνει τη συγγήτριά μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Νταφ. Ο κύριος Χέφνερ. Ναι, <clears throat> πρώτα απ' όλα ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια και την πολλή δουλειά που έκανε βήμα προς τα εμπρός το ότι μιλάμε για ξεκάθαρες διαφανείς ε, δημοκρατικές διαδικασίες και κανόνες. Είχαμε μία δυστυχώς ε, μία φοβερή ε, ακρόαση. Φοβάμαι πως δυστυχώς πρέπει να ασκήσω κάποια κριτική γιατί πάρα πολλά από αυτά τα οποία είχαμε πει στο σχέδιο έκθεσης λυπούμε γιατί βλέπω πως δεν ε, περιέχονται εδώ πέρα. Θέλω να αναφέρω ένα αποφασιστικό ζήτημα. Η σχέση της αναγνώρισης και χρηματοδότησης των κομμάτων η οποία αντιμετωπίζεται ως κάτι το ενιαίο στην έκθεση. Να σας πω κάτι. Εγώ ο ίδιος πριν από 33 χρόνια ίδρυσα ένα κόμμα το οποίο δεν υπήρχε πριν. Δηλαδή ήταν ένα κόμμα για το οποίο δεν υπήρχε κάποια πρόδρομη οργάνωση ή κάτι τέτοιο. Ήταν ένα κόμμα το οποίο τη στιγμή της ίδρυσης δεν εκπροσωπούταν δεν εκπροσωπούνταν πουθενά σε κανένα κοινοβούλιο γιατί δεν υπήρχε. Του δώσαμε το όνομα Πράσινη και σήμερα είμαστε σε πολλά κοινοβούλια, είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, σε κυβερνήσεις και τα λοιπά και είναι λογικό για τη δημοκρατία να έχουν την ε, ευκαιρία οι νέες οργανώσεις και τα κόμματα να ε, μπουν σε αυτόν τον δημοκρατικό ανταγωνισμό. Γιατί σκεφτείτε ε, τον κίνδυνο που υπάρχει αν κάνουμε πολιτική προς το συμφέρον μας και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή γιατί όλοι είμαστε μέλη πολιτικών κομμάτων και θα έπρεπε να αποφύγουμε αυτά τα οποία κάνουμε τώρα να είναι προς το συμφέρον των δικών μας κομμάτων τόσο ώστε να περιορίζουμε αντί να ανοίγουμε τον ανταγωνισμό. Οπότε η αδειοδότηση, αναγνώριση, όλα αυτά των πολιτικών κομμάτων δεν μπορούν να συνδεθούν με την εκλογική επιτυχία. Δεν μπορούν να συνδεθούν με το να βρίσκεται ήδη σε κάποιο κοινοβούλιο το κόμμα. Αυτό είναι τελείως αντίθετο με την ιδέα του ελεύθερου ανταγωνισμού σε μια δημοκρατία. Και δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Αλλιώ έχουν τα πράγματα με την χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση πρέπει να συνδέεται με ένα κριτήριο επιτυχίας. Εκεί πέρα είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο ε, λέει η έκθεση και θα μπορούσαμε να θέσουμε και αυστηρότερα κριτήρια, αλλά όσον αφορά την αναγνώριση και το να το ταυτίζει δηλαδή, ε, είναι κάτι το, το απαράδεκτο. Οπότε, κυρία Γιαννάκου, η συμβιβαστική τροπολογία που αγγίζει αυτό το θέμα για τις, ε, όπου έχετε θέσει ως όρο χρηματοδότησης ε, την εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ξεκαθαρίζει τα πράγματα γιατί εξακολουθεί να παραμένουν ε, οι προϋποθέσεις αυτές αναγνώρισης ε, να παραμένουν ασαφείς. Πρέπει να, δεν μπορεί να το συνδέουμε με την επιτυχία, πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα, πρέπει να υπάρχει ένας επαρκής αριθμός μελών, να υπάρχει εσωτερική δημοκρατία, ένας επαρκής αριθμός υποστηρικτών κτλ. Ένα καταστατικό ένα καταστατικό το οποίο θα διασφαλίζει πως οι αποφασίσεις ε, εντός του κόμματος λαμβάνονται δημοκρατικά κτλ. Αλλά δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να συνδέεται με ήδη ε, εκπροσώπηση σε προηγούμενες εκλογές. Αλλιώς κάνουμε εδώ πέρα ένα ολιγοπόλιο των ε, υπαρχόντων ήδη και δεν είναι σωστό. Οπότε θα ήθελα να σα παρακαλέσω να το ξαναδείτε αυτό, να το επανεξετάσετε. Και να δείτε και τις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει σχετικά. Και να σα υπενθυμίσω πως είχα αναφέρει κάτι τέτοιο και στην ακρόαση και όλοι όσοι αναφέρθηκαν μετά από μένα στο ίδιο ζήτημα ανέφεραν ακριβώς το ίδιο σημείο. Όλοι οι ειδικοί που μίλησαν είχαν ακριβώς την ίδια θέση. Οπότε Ήθελα να θέσω εδώ πέρα το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων και απευθύνω έκκληση να αποφύγουμε τον κίνδυνο να κάνουμε πολιτική προς το δικό μας ε, συμφέρον και να μην, ε, να μην δημιουργήσουμε αυτό το ολιγοπόλιο το οποίο δεν θα εξυπηρετήσει την ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτά έχετε δει και τις υπόλοιπες ε, τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Τρεις συναδέλφους ε, βλέπω στον κατάλογο των ομιλητών. Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα ήθελε να αναλάβει το λόγο. Όχι, κυρία Μαντάμ Λεκρύπ, λοιπόν. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την συγγήτριά μας, την κυρία Γιαννάκου. Συγχαρητήρια, κυρία Γιαννάκου. Ε, ήταν Ηράκλειο το έργο σας ε, και τώρα περατώνεται μετά από, αν κατάλαβα καλά, μετά από μια μακρά διαδικασία που ξεκίνησε στην προηγούμενη θητεία, αλλά εν πάση περιπτώσει φτάνει ε, σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο η διαδικασία και θα περατωθεί όπως έλεγα. Ε, συγχαρητήρια και για τα αποτελέσματα της ακρόασης που έλαβε χώρα στα τέλη Ιανουαρίου. Όλα τα κόμματα εκπροσωπήθηκαν και τα περισσότερα σε ανώτατο επίπεδο. Αυτό καταδεικνύει το ενδιαφέρον που παρουσίαζε η ακρόαση και ε, ο, καταδεικνύει επίση ότι ε, χειρίστηκε με επιδέξιο τρόπο η Επιτροπή το ζήτημα. Η συνθήκη της Λισαβόνας επίσημα αναγνωρίζεται ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα το ρόλο τους, ε, τη σημασία της ε, συνεισφοράς τους ε, για την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου και τη συμβολή τους στην ανάδειξη μιας ευρωπαϊκής κοινή γνώμης, ούτως ώστε να υπάρχουν πραγματικά ευρωπαϊκοί διάλογοι, ανταλλαγή απόψεων και όπως και η ευρωπαϊκή ηθαγένεια εξάλλου, ο στόχος ε, που επιδιώκουμε είναι αυτό συγκεκριμένα να εμπλακούν στα κοινά οι πολίτες της Ένωσης. Βέβαια οι σοβαρότατοι πολιτικοί κλειδονισμοί που ε, βιώνουν οι άνθρωποι από την άλλη πλευρά της λεκάνης της Μεσογείου μας ε, δείχνουν ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε στα χέρια μας το κατάλληλο εργαλείο, το κατάλληλο μέσο για να συνοδεύσουμε τις ε, δημοκρατικές διαδικασίες, τα πολιτικά κινήματα που αγγίζουν ε, την Εγγύς και τη Μέση Ανατολή είναι σημαντικό για στα κάθε μας και κατά τη διάρκεια των εκλογικών διαδικασιών που μας ενδιαφέρουν πρωτίστως να ε, διαδραματίσει το διάλογο ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτως και γι' αυτό χρειαζόμαστε μία ενιαία αναγνώριση, ένα κοινό πλαίσιο, ένα κοινό νομικό καθεστώς για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Θα ήθελα μόνο να διευκρινίσω πριν κλείσω από τις ε, τροπολογίες ε, που υποβάλαμε από κοινού με τον κύριο Λαμασούχ ε, για το φορολογικό καθεστώς του προσωπικού των πολιτικών ομάδων. Δύο τροπολογίες που προτείνουν την κατάργηση του εκτιμώντας τη λογική σκέψη ΑΑ ένα αλφα συγγνώμη, και της παραγράφου 10 που αναφέρεται στο φορολογικό καθεστώς του προσωπικού των κομμάτων εκφράζουμε την αμηχανία μας, ε, την ε, ε, έλλειψη κατανόησης για ένα ιονίδιο ενιαίο φορολογικό καθεστώς ε, για τα κόμματα, δηλαδή θα ευθυγραμμιστούν όλοι από φορολογική πλευράς ε, με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη. Ή να φανταστούμε ένα ad hoc ε, φορολογικό καθεστώς, θεωρώ ότι σε αυτό το στάδιο ακόμη δεν έχουν αποκρισταλωθεί οι απόψεις μας για αυτό το ζήτημα ζήτημα, αλλά πάντως εκφράζουμε την έλλειψη κατανόηση από πλευρά μας μέσα στις τροπολογίες μας και ταυτόχρονα θέλουμε να περάσουμε το εξής μήνυμα. Ένα τέτοιο φορολογικό καθεστώς θα έπρεπε να συζητηθεί ευρέως, ε, να εμβαθύνουμε στην εξέταση αυτού του ζητήματος πολλές πολιτικές ομάδες εξέφρασαν αυτήν την ε, ε, επιθυμία ε, πάντως θεωρώ ότι δεν είναι όριμο αυτό το θέμα, το αντίθετο οδηγεί σε έλλειψη κατανόησης και σε ενδιασμούς, σε αμφιβολίες ε, για πολλούς από μας και για πολλούς από τους συμπολίτες μας. Ε, αυτά σχετικά με το ρόλο των ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής διαδικασίας. Αυτά τα ζητήματα, ε, ξέρετε, ενδιαφέρουν άμεσα πολλούς συμπατριώτες μας, πολλούς συμπολίτες μας. Εγώ ε, συχνά ακούω από νέους συμπολίτες μας ότι ναι, επιθυμούν το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα να είναι πιο ενεργό, να δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή σκηνή περισσότερο αλλά προς Θεού ας μην περιπλέξουμε την υπόθεση γιατί αυτό το ακαθόδε ζήτημα καλό είναι να εξεταστεί με γενέστερα. Με αυτές λοιπόν μόνο τις αμφιβολίες, με αυτούς τους ενδιασμούς ε, επικροτώ και πάλι τους καρπούς των εργασιών σας ε, κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστούμε Κωνσταντς ο κύριος Σόλτς, Μπρόγκς ε, και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος, αλλιώς να κλείσουμε τον κατάλογο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που ευχαρίστησαν την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει γίνει και για την πολύ επιτυχημένη ακρόαση. Αυτό το οποίο προέκυψε θεωρώ από την ακρόαση ήταν πως όλα τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γνωρίζουν πως πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός εάν θέλουμε να έχουμε πιο δημοκρατική συμμετοχή πολιτών και μεγαλύτερη πολιτική υπευθυνότητα των κομμάτων. Ο Βρετανός κοινωνιολόγος Colin Crouch ε, μίλησε κάποτε για την μεταδημοκρατία στο πλαίσιο του ότι όλο και λιγότεροι πολίτες συμμετέχουν πλέον στις εκλογές παρά το ότι έχουν τα κράτη-μέλη της Ένωσης ε, δημοκρατικούς θεσμούς, ελεύθερες εκλογές, ε, ελευθερία γνώμης κτλ. Δηλαδή δεν θεωρούν πως τους αγγίζει η διαδικασία λήψη αποφάσεων στην πολιτική. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα πολιτικά κόμματα και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και προέκυψε αυτό και στην ακρόαση πως ε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κάποιον έτσι πανευρωπαϊκό χαρακτήρα των κομμάτων. Τώρα, για την έκθεση και τις συμβαστικές τροπολογίες που έχουμε μπροστά μας, θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία θέματα τα οποία είναι για εμάς σημαντικά. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Έθνερ όσον αφορά τον διαχωρισμό μεταξύ ε, αναγνώρισης και χρηματοδότησης. Είναι πολιτικά κόμματα όπως τα γνωρίζουμε στην καθημερινή δημοκρατική καθημερινότητα, στην καθημερινή ζωή της δημοκρατικής κοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κάποιες οργανωτικές αρχές που θα πρέπει να είναι η προϋπόθεση για αναγνώριση από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεύτερον για το ζήτημα της χρηματοδότησης, ε, εκεί πέρα συμφωνώ πάλι με τον συνάδελφο, εκεί πέρα μπορούμε να έχουμε το κριτήριο της εκλογικής επιτυχίας. Ο, βεβαίως, όπως προσπάθησα να ξεκαθαρίσω και σε μια τροπολογία, οι υπάρξεις ρυθμίσεις που έχουμε από το 2007 για εμένα επαρκούν. Και αυτό βεβαίως αφορά και το ζήτημα των ερετών μελών σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο που μπορούν να είναι σημαντικά για ένα κόμμα γιατί έτσι γίνεται σαφές πως το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα δεν είναι κάτι το αφηρημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά πρέπει να συνδέεται με την πολιτική ζωή των μελών στα κράτη-μέλη με τα εθνικά κόμματα και έτσι να προωθηθεί η ευρωπαϊκή διαδικασία Διαμόρφωση της γνώμη. Γι' αυτό είναι σημαντικό, επειδή σπάμε το κεφάλι μας, το τι θα, το τι θα συνεισφέρει ε, το ευρωπαϊκό αυτό κόμμα, δηλαδή αν θα κάνει προεκλογικές εκστρατείες και τα λεπά. Κατόπιν και τις πολλές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για την δημοκρατία κτλ. Θεωρώ πως θα πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες και όσο, όσες απαιτούνται ε, περιορισμούς. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι σε θέση τα μέλη του εκάστοτε κόμματο να διαμορφώνουν από μόνοι του και του κανονισμού και βεβαίω την γνώμη του εντό του κόμματο με βάση κάποιε απλέ και βασικές αρχές βεβαίως που θα οριστούν. Και εδώ πέρα βεβαίως κατά την άποψή μου ανήκει και η δυνατότητα της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής στις εργασίες των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και εκεί πέρα δηλαδή να γίνει το κατόφλιο στο δυνατόν πιο χαμηλό. Τρίτον, για τα μέλη και πάλι, και εκεί πέρα έχω καταθέσει κάποιες ε, τροπολογίες μαζί με άλλους ε, και άλλοι συναδελφοί. Θεωρώ πως και τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη εδώ πέρα. Να μπορούν να είναι μέλη Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος γιατί ακριβώς αυτή είναι η παραπάνω ιδιότητα που έχει το Ευρωπαϊκό ε, Πολιτικό Κόμμα. Βεβαίως υπάρχει και η συμβαστική λύση η οποία προτάθηκε στο νέο άρθρο 3, στην παρά, άρθρο 9 παράγραφος 31 ε, όπου ζητάμε να δούμε ποια θα είναι η σχέση μεταξύ μεμονωμένων μελών και άμεσης συμμετοχής ε, των μελών και των συλλογικών μελών, δηλαδή των ιδίων των κομμάτων στα ευρωπαϊκά κόμματα. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα πτυχή και νομίζω πως μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη συμβαστική λύση εδώ πέρα. Να πω επίσης, τέλος, πως και ο ρόλος των πολιτικών ιδρυμάτων των νέων και ειδικά των δομών των γυναικών ε, στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Θα πρέπει να είναι δομές που θα δίνουν, την, θα δίνουν περισσότερες δυνατότητες στο ευρωπαϊκό επίπεδο στην άμεση διαμόρφωση γνώμης όσον αφορά την, ε, την ευρωπαϊκή πολιτική. Και από εκεί άρα θα οδηγηθούμε ίσως ε, δεν ξέρω και εισάτοπον με αυτή τη μεταδημοκρατία που είχε πει και ο Άγγλος ε, κοινωνιολόγος και εδώ πέρα θα ήθελα να συμφωνήσω με τον ε, Άντριου Νταφ Ευχαριστώ κύριος Μπρόντς Is it ε, Ωραία. Λειτουργεί. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα υπάρχουν μόνο ως ομπρέλες, συμμαχίες εθνικών κομμάτων. Αλλά βέβαια η βασική λειτουργία ενός πολιτικού κόμματος είναι να κατεβαίνει στις εκλογές. Και από όσο ξέρω οι συμμαχίες αυτές δεν κατεβαίνουν στις εκλογές. Ε, υπό το ενιαίο τους όνομα πουθενά στην Ευρώπη. Η μόνη δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο είναι εάν περάσει η πρόταση DAF ε, περί Ευρωπαϊκής Περιφέρειας 25 Ευρωβουλευτών. Και πάλι βεβαίως θα μιλάμε για μικρή μειοψηφία του συνολικού αριθμού Ευρωβουλευτών. Δεν πιστεύω πως οποιοδήποτε εθνικό πολιτικό κόμμα ανεξάρτητα και αυτοβούλος και αυτόνομα θα κατέβει στις εκλογές ε, ε, υπό ένα άγνωστο όνομα Ευρωπαϊκού Κόμματος. Αυτό θα είναι εκλογική αυτοκτονία, κατά το οποίο βεβαίως υποδηλώνει πως δεν θα κατέβουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα σε εκλογές αυτοβούλος. Οπότε, αν συνεχιστεί αυτό, τότε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα είναι πειραματικά και πολύ ακριβά παρανθετικά και ε, πολύ ακριβά πρωτότυπα, εάν θέλετε. Η μόνη, ε, ο μόνος τρόπος βεβαίως για να κατέβουν ε, στις ε, εκλογές είναι το να γίνουν υποχρεωτικά, κατά το οποίο νομίζω πάει πάρα πολύ μακριά τα και να απαγορεύσουμε τα εθνικά κόμματα. Η ιδέα η οποία προτάθηκε είναι πως κάποιοι θα θέλουν να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα νομίζω ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Είμαστε δηλαδή σε θέση να συζητάμε λεπτομερείς κανόνες για πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στον πραγματικό κόσμο. Υπάρχουν εδώ πέρα, τα γνωρίζουμε εμείς, αλλά δεν τα γνωρίζει ο πολλής κόσμος. Εάν κάνετε μια δημοσκόπηση στα κράτη-μέλη για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, θα σας κοιτούσαν και δεν θα ήξεραν τίποτα. Οπότε τι κάνουμε, συζητάμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει, δεν το ξέρουν οι περισσότεροι άνθρωποι και δεν θα υπάρξει στην βασική λειτουργία του να κατεβαίνει σε ευρωεκλογές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλώ. Νομίζω ότι η η ώρα τη απάντηση από πλευρά της εισηγήτρια, η οποία θα μπορούσε ίσω να μα παρουσιάσει και τι συμβαστικέ τροπολογίε που άκουσα. Παρακαλώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, άκουσα τις παρατηρήσεις όλων των συναδέλφων. Ε, βρίσκω ότι κατά βάση αυτό στο οποίο έχουν αντίρρηση είναι ένα European ε, legal and fiscal status για, το staff και το καταλαβαίνω ότι ίσως θα ισχυριζόταν κανείς ότι δεν είναι του παρόντος. Βέβαια, εγώ δεν είχα στο νου μου ένα στάτους ίδιο με, το, με τους φονξιονέα, με τους υπαλλήλους, ούτε με τους βοηθούς. Εννοούσα ένα ad hoc στάτους. καταλαβαίνετε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, δεν είναι το μείζον θέμα. Το μείζον θέμα είναι να υπάρχει ε, ένα political, legal ε, και λοιπά στάτους για τα κόμματα και, τις, ε, και τα ιδρύματά τους και επίσης να ξεκαθαρίσουμε <clears throat> ότι αυτή τη στιγμή βεβαίως σημειώνεται στην παράγραφο 31 ότι μπορούν να είναι και μέλη, δηλαδή να συμμετέχουν πρόσωπα στα κόμματα αυτά, αλλά για να δημιουργηθούν ευρωπαϊκά κόμματα και να έχουν μεγάλο αριθμό προσώπων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό χρειάζεται πάρα πολλά χρόνια, πολύ χρόνο. Ε, υπάρχει, υπάρχουν τροπολογίες συμβιβαστικές στις οποίες γίνεται αποδεκτή η έννοια της διαφοροποίησης ανάμεσα στα κόμματα και σε αυτά που χρηματοδοτούνται. Γιατί είδα ότι όλοι ε, ζήτησαν για να χρηματοδοτούνται να έχουν τουλάχιστον ένα μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό είναι λογικό. Και εγώ δεν έχω διαφωνία, υπάρχει η τροπολογία η συμβιβαστική, δεν διαφωνώ να αναγνωρίζετε το στάτους των κομμάτων ε, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν πριν από εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και βεβαίως εάν εκλέξουν ε, μέλη να χρηματοδοτούνται. Ε, επίσης για μένα ευαίσθητο είναι το σημείο της χρηματοδότησης. Αυτή τη στιγμή ακόμα και αν εγγράψουν πολλά μέλη δεν είναι αρκετά τα χρήματα αυτά για να μπορούν να σταθούν. Καταλαβαίνετε ότι τα μέλη πληρώνουν αυτή τη στιγμή στα περισσότερα κόμματα 20 ευρώ το χρόνο. Επομένως και αυτό είναι μελλοντικό. Θα πρέπει η χρηματοδότηση να παραμείνει έτσι. Θέλω να σημειώσω ότι από τη συζήτηση που έκανα με όλα τα κόμματα δεν ζητούν περισσότερα χρήματα. Γιατί πράγματι αντιλαμβάνομαι η εποχή είναι ευαίσθητη, υπάρχει οικονομική κρίση, η κριτική που γίνεται στους πολιτικούς και στα κόμματα είναι πολύ έντονη και από τα μίντια και από τους πολίτες ε, όμως η προσπάθεια αυτή για τα κόμματα είναι κάτι που εντάσσεται και πολύ σωστά υπόθηκε ε, σε όλες τις προσπάθειες που κάναμε και μέσα στη συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης δηλαδή ε, μεγαλύτερη επαφή με τους πολίτες η πρωτοβουλία των πολιτών να γνωρίσουν οι πολίτες τι σημαίνει Ευρωπαϊκό Κόμμα σε ορισμένες χώρες γνωρίζουν τα ευρωπαϊκά κόμματα γιατί έχουν δραστηριότητες μαζί με τα εθνικά κόμματα. Είναι μια προσπάθεια δηλαδή προσέγγισης των πολιτών, εκδημοκρατισμού, διαφάνειας και εφόσον έχουμε μια ένωση με μια νομική προσωπικότητα, εφόσον έχουμε ελεύθερη διακίνηση αγαθών προσώπων υπηρεσιών κεφαλαίων, εφόσον βασικά ζητήματα της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής ελέγχονται σε επίπεδο θεσμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι είναι πάρα πολύ φυσικό να ενισχύσουμε όσο μπορούμε την έννοια του ε, κόμματος. Από τις παρατηρήσεις αυτές που έγιναν ε, σας τόνισα το θέμα της διάκρισης από τον κύριο Γκερέρο και τον κύριο Νταφ σημειώνω ε, αυτή του κυρίου Νταφ για την πιο σκληρή πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί και από εμά, δεν είναι μόνο η έκθεση. Θα πρέπει ίσως η Επιτροπή και αν συμφωνεί ομόφωνα να αποστείλει και μια, ένα επίσημο, μια επίσημη επιστολή στην Επιτροπή η οποία θα πρέπει να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες για να φέρει μια πρόταση. Και νομίζω ότι ο χρόνος ε, έχει επέλθει. Τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν μπορούν να βρεθούν άλλες δικαιολογίε. Ε, και βέβαια ε, ελέγχθη κάτι για, για πολιτική ιδίου συμφέροντος για τα χρηματοδότηση. Εγώ δέχομαι τη σοσιαλιστική τροπολογία, την έχω εντάξει μέσα σε συμβιβαστική τροπολογία, 25.000 ευρώ ανά πρόσωπο και ανά έτος. Νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που είπατε κύριε Γκερέρο και είναι και λογικό και βεβαίως ε, όπως αντιλαμβάνεστε κάτω από συνθήκες ε, κανόνων και συγκεκριμένου καθεστώτος των κομμάτων είναι φυσικό να υπάρχει και μεγαλύτερη διαφάνεια και να μπορούν να ελέγχονται πολύ καλύτερα τα οικονομικά τους. Ε, οι τροπολογίες που έχω κάνει δεν είναι μεγάλες, έχουν σκοπό να μειώσουν κατά κάποιο τρόπο γιατί υπάρχουν και 99 τροπολογίες. Όπως σας είπα λοιπόν στην αρχή, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ελεύθερη ψηφοφορία στο θέμα του στάτους του ΣΤΑΦ. Ε, θέλω να επιμείνω και να σας παρακαλέσω να ψηφίσετε το κομμάτι το οικονομικό, έτσι όπως έχω αποδεχθεί την τροπολογία του κυρίου Γκερέρο και ε, συνδυάζεται με το ποσοστό που δίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί δεν είναι του παρόντος ε, να μαζεύει μόνο του ένα Ευρωπαϊκό Κόμμα τα χρήματα, πρέπει να αρχίσει να γράφει μέλη και μετά χρειάζεται χρόνος για αυτό το πράγμα. Ε, και βεβαίως η απέτησή μας πρέπει να είναι για ένα στάτους των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων σε πολιτικό, νομικό και φορολογικό επίπεδο. Τα κόμματα και βέβαια και τα ιδρύματά τους και σημειώνω στην έκθεση τα ιδρύματά τους διότι ε, αυτά είναι ιδρύματα που συνδέονται με τα συγκεκριμένα κόμματα. Τα ιδρύματα χρηματοδοτούνται λόγω της χρηματοδότησης των κομμάτων. Δεν χρηματοδοτούνται αυτονόμως. Δηλαδή, εάν εμφανιστεί αύριο ένα ίδρυμα και πει ότι είναι ίδρυμα σοσιαλιστικού χαρακτήρα, αυτομάτως θα τεθεί δίπλα στη Σοσιαλιστικό Κόμμα. Όχι. Θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτό Επομένως είναι σωστό και το affiliated που περιλαμβάνεται στις κυρία Γκουρμάη την τροπολογία το οποίο εγώ ε, επιλύω με μια τροπολογία συμβαστική η οποία μνημονεύει το συγκεκριμένο άρθρο, τη συγκεκριμένη παράγραφο και όπως ακριβώς αναφέρεται στον κανονισμό όπου έτσι ακριβώς αναφέρονται δηλαδή European Parties and their affiliated foundations και νομίζω ότι εκεί ε, μπορούμε να μείνουμε σύμφωνοι. Ε, κύριε Πρόεδρε, εγώ έκανα την μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια. Πολλά, πολλές τροπολογίες είναι παρόμοιες ε, ή και ίδιες τελείως μέσω των συμβαστικών αυτών τροπολογιών ώστε να καλυφθεί μεγάλο μέρος των τροπολογιών και να μην καταστραφεί ο πυρήνας της έκθεσης που είναι η βούλησή μας να αποκτήσουν πραγματικό καταστατικό με νομικό χαρακτήρα τα ευρωπαϊκά κόμματα και ε, τα ιδρύματά τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Γιαννάκου. Σας ευχαριστώ ειλικρινά και για την εκθεσή σας και για την απάντησή σας. Να περάσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερησία διάταξη για σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, ποιος θέλει να μιλήσει, παρακαλώ, ο κύριος Χέφνερ. Δεν σας είχα δει. Έχω, μια παράκληση. Πριν να τελειώσουμε με αυτό το θέμα, θα ήθελα να ρωτήσω την εισηγήτρια μήπως θα μπορούσε να απαντήσει και στο ερώτημα το δικό μου. Ε, έκανα μία μόνο ερώτηση γιατί θεωρώ πως ε, θα πρέπει ε, να δούμε ειδικά το ζήτημα το οποίο αφορά την δική μας ε, την Επιτροπή των Συνταγματικών Θεμάτων και ε, με εξέπληξε το ότι δεν, δεν απαντήθηκε αυτό το ερώτημα. Νομίζω εξαρτάται η... θα εξαρτηθεί η στάση μας από το πώς θα, θα απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση, οπότε θα ήθελα σας παρακαλώ να απαντήσετε. Μπορείτε. Σα υπενθυμίζω την ερώτηση. Μπορείτε να απαντήσετε. Θέλετε να απαντήσετε, κυρία Γεννάκου, στον κύριο Χέφνερ. Ε, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Χέφνερ έκανε μια ερώτηση για τη διάκριση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κόμματος και της χρηματοδότησής του. Και είπα ότι μέσω της, ε, των τροπολογιών των συμβαστικών αυτό αναγνωρίζεται. Δεν υπάρχει στην έκθεση, αλλά αναγνωρίζεται μέσω των συμβαστικών τροπολογιών. Και είπα ότι συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξουν κριτήρια αναγνώρισης, βέβαια δεν μπορούν να αναφέρονται εδώ. Εδώ αναφέρεται το κριτήριο της χρηματοδότησης, που είναι η εκλογή ενός Ευρωπαίου βουλευτή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κόμματα που θα δημιουργηθούν πριν από ευρωπαϊκές εκλογές δεν μπορούν να αναγνωρίζονται ως ευρωπαϊκά κόμματα και μέχρι ότου βεβαίως ε, εκτεθούν και σε εκλογές αλλά εν πάση περιπτώσει εφόσον εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις διότι δεν μπορούν να αγνοήσουν τα ευρωπαϊκά κόμματα ε, τα κόμματα μέλη δηλαδή δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ούτε την εγγραφή στα ευρωπαϊκά κόμματα προσώπων ούτε τα κόμματα μέλη. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ένας συνδυασμός κομμάτων και κομμάτων μελών. Από εκεί και πέρα θα έρθει μια πρόταση και αυτό θα αναγνωριστεί. Τώρα αυτό θα μπορούσε να μπει και σε μια εξτρεμιστική λογική, δηλαδή μια ομάδα πέντε ανθρώπων να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό κόμμα χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, χωρίς κόμματα μέλη, χωρίς τίποτα. Ε, αυτό κύριε Πρόεδρε δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρείται ευρωπαϊκό κόμμα. Αυτό είναι σαφές. Επομένως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να είναι ευρωπαϊκό κόμμα κάποιο και υπάρχει και η βασική προϋπόθεση για να χρηματοδοτείτε. Äh, για να επανέλθω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γεννακού, με άλλη μια ερώτηση. Αν μπορείτε να δεχτείτε την, ε, την πρόταση αυτή που που αναφέρατε τώρα προφορικά και σας ευχαριστώ γιατί δεν υπάρχει μέχρι στιγμή ούτε στην έκθεση ούτε, ούτε στις συμβαστικές τροπολογίες. Αλλά εάν κάνετε αυτά τα οποία μας είπατε τότε νομίζω ότι έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και μπορούμε να έχουμε μια λύση. Ωραία. Ευχαριστώ. Ακούσατε και την απάντησή σας και από εκεί και πέρα θα δείτε τι στάση θα κρατήσετε. Να περάσουμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 8, ερμηνεία του άρθρου 51, κοινέ συνεδριάσει επιτροπών. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί το έχουμε ήδη συζητήσει το θέμα αυτό στη συνεδρίαση της 31 Ιανουαρίου και σας έχει διανεμηθεί και ένα σχέδιο έκθεση τροποποιημένο να σας πω ότι στην τελευταία συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων, στις 8, των Προέδρων Επιτροπών, στις 8 Μαρτίου, είχα παρουσιάσει και το συγκεκριμένο θέμα. Θα θυμάστε ότι η έκθεσή μου προκύπτει από μια ερώτηση που έθεσε ο, Επιτροπής, ο Πρόεδρος Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων που ζητούσε εναλλακτικέ λύσεις και ήθελε να ξέρει τι σχέση υπάρχει μεταξύ των άρθρων 50 και 51 και πιο συγκεκριμένα η διαδικασία του άρθρου 51 ισχύει για όλη την νομοθετική διαδικασία ή μόνο για την πρώτη ανάγνωση. Δεύτερον, η Η Δευτερεύουσα Επιτροπή έχει όλα τα δικαιώματα με ε, την αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή ε, και μπορεί για παράδειγμα να αποσύρει και την ε, νομοθεσία που παρουσιάζεται. Και τέλος, κατά πόσον η κοινή διαδικασία ισχύει και για τις ε, εκτελεστικές πράξεις και τις πράξεις εξουσιοδότηση. Εμείς σας απαντήσαμε σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις και είπαμε ότι σαφώς ε, θα πρέπει, αυτή τη έχει καθοριστεί ότι θα εφαρμοστεί το άρθρο 51, δηλαδή η κοινή ε, διαδικασία ισχύει για όλη την ε, νομοθετική διαδικασία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής προϋπόθεση που κάνει και τη διάκριση μεταξύ των άρθρων 50 και 51 και θεωρεί έκτακτη τη χρήση του άρθρου 51. Και αυτό είναι το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό να διακρίνουμε ποια, ε, ποιο θέμα είναι αρμοδιότητας ποιας επιτροπής και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε κοινή αρμοδιότητα. Το καλύτερο θα ήταν να εφαρμόζεται το άρθρο 50, αλλά αν δεν μπορεί να γίνει η διάκριση, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 51. Ούτω ή άλλω πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο και το θέμα όμω είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν μιλάμε για θέματα δευτερευούση σημασία, δεν υπάρχει λόγο να περιπλέξουμε τόσο πολύ τα πράγματα. Ακόμα και αν είναι αρμόδια μία επιτροπή η οποία θα πρέπει ίσως να ασχοληθεί και με θέματα τα οποία δεν είναι τόσο της ε, αρμοδιότητάς της, δεν είναι και πολύ σημαντικό το πρόβλημα εάν είναι δευτερευούση η στα ζητήματα αυτά. Τώρα, ο πρόεδρος ε, Λένε έχει ζητήσει να ε, απλουστεύσουμε τη διαδικασία στην παράγραφο 4 και η παράγραφος 4 ε, με δική μου τροπολογία προβλέπει οι δύο επιτροπές οι οποίες θα δρούν από κοινού όταν ε, αποφασίζεται η χρήση του άρθρου 51 μέχρι την εκτελεστική διαδικασία και στην εκτελεστική διαδικασία η διάκτηση σκέψη των Προέδρων μπορεί να επιλέξει μία εκ των δύο επιτροπών. Και στη διάσκεψη των Προέδρων προτείνεται να βρεθεί ένα μηχανισμό που να μα επιτρέψει να δράσουμε πιο γρήγορα και θα προσπαθήσουμε να δούμε πώ μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι θα παρουσιάσω και τροπολογία επί του θέματο. Η δεύτερη παρατήρηση που έγινε από τον πρόεδρο Λάινεν τη Επιτροπή περιβάλλοντο, είναι να υπάρχουν κάποιε προθεσμίε για τι συνεδριάσει των κοινών επιτροπών στη δεύτερη ανάγνωση, γιατί αλλιώ ελοχεύει ο κίνδυνο να μην μπορούμε να σεβαστούμε τα χρονοδιαγράμματα και επομένω θα έπρεπε να δούμε κατά πόσον είναι δυνατή και νομίζω ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε μια τροπολογία που θα επιλύει το σχετικό πρόβλημα. Τώρα, να περάσουμε στη συζήτηση. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 15 Μαρτίου, αύριο δηλαδή το βράδυ τα μεσάνυχτα. Ο συνάδελφος Γκερέρο όμως ζητά παράταση για την κατάθεση των τροπολογιών. Προτείνω να σας δώσω μέχρι τις 24 Μαρτίου τις τροπολογίες τις οποίες θεωρώ ότι θα πρέπει να παρουσιάσω και σας παρουσίασα και το ανακοίνωσα τώρα και να αλλάξουμε λοιπόν τα πράγματα και να βάλουμε γενική προθεσμία των τροπολογιών της, την Πέμπτη για να έχουμε χρόνο να, να παρουσιάσουμε τις τροπολογίες. Αν συμφωνείτε μου το λέτε. Ο κύριος Βίλαντ έχει ζητήσει το λόγο. Ναι, δύο σύντομες παρατηρήσεις. Η πρώτη το ότι λέμε πως αυτό το θέμα έχει μεγάλη σημασία. Αυτό είναι κάτι το, το υποκειμενικό. Και δεύτερον, πως το ζήτημα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, ο καθένα εδώ μέσα όποιο θέμα ασχολείται, με όποιο θέμα ασχολείται, το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι τόσο υποκειμενικό το κείμενο αυτό εδώ πέρα και έχει τέτοιους όρους ώστε θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, όταν μιλάμε για ζητήματα αρχής που αφορούν τις επιτροπές, γιατί αυτό το θέμα που για μένα είναι οργανωτικό ε, ζήτημα και ζήτημα αποτελεσματικότητας γιατί είναι αρμοδιότητας διάσκεψης των προέδρων και, των, και όχι της διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών. Και κάτι άλλο. Στο σημείο 11 έχουμε την έκθεση DAF που αφορά την ακρόαση της Κομισιόν και εκεί πέρα μιλάμε ξαφνικά για συνδεδεμένες επιτροπές συνεχώς εφευρίσκουμε νέα μέσα. Κάποια στιγμή χρησιμο... θα... εδώ πέρα θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη μικτές επιτροπές και βεβαίως στο, στο έργο του κυρίου Κασίνη θα έπρεπε να μιλάμε για κοινέ ακροάσεις ε, επιτρόπων που καλύπτουν περισσότερες επιτροπές. για να δημιουργηθεί έτσι και ένας ε, κανόνας ο οποίος ε, θα, εφαρμόζεται κάθε πέντε χρόνια. Για να γίνει έτσι λίγο πιο λογική όλη η διαδικασία. Κύριε Κυρέρο, καταρχάς ε, ζητώ συγγνώμη γιατί παρεμβαίνω σε όλα τα σημεία της συζήτησης σήμερα. Μάλλον είμαι η ξεχωριστή περίπτωση που ανέφερε ο κύριο Βίλαντ υπό την έννοια ότι επειδή έχω άποψη παντό επιστητού κατά πάσα πιθανότητα δεν λέω και τίποτα σημαντικό. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια παρεμβαίνω εξ ονόματο στον Ντέιβιτ Μάρτιν που είναι ο σκιώδης εισηγητής ε, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και θα ήθελα να σας πω ότι Κατά την άποψή μας αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η διαδικασία αυτή να χρησιμοποιείται το λιγότερο δυνατόν. Και όταν η διάσκεψη των Προέδρων ε, των Επιτροπών αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία, θα είναι σαφές ότι πρόκειται για αρμοδιότητες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες ε, και είναι σχεδόν εξίσου τις αρμοδιότητες και των δύο περισσότερων ε, επιτροπών και είναι θέμα μείζων σημασία. Αυτό που αναφέρεται στα αγγλικά, major importance, θα πρέπει να γίνεται σεβαστό, να ακολουθούμε πιστά τη διατύπωση. Τα προβλήματα που προκύπτουν, επειδή σε γενικές γραμμές ε, συμφωνούμε με το πνεύμα της έκθεσης του κύριου Καζίνη. Τα προβλήματα λοιπόν που τίθενται αφορούν τη χρήση του χρόνου, δηλαδή τα προβλήματα που μπορούμε να έχουμε από χρονική σκοπιά και το το διαφορετικό μέγεθος των επιτροπών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στη διαδικασία. Όσον αφορά τη χρονική πτυχή, θεωρούμε ότι η εσωτερική μάχη μεταξύ διαφορετικών επιτροπών για την ενασχόλησή τους με ένα θέμα ή η καθυστέρηση της διάσκεψης των Προέδρων να λάβει απόφαση επί του θέματος μπορεί να μας οδηγήσει στο εξή. Να περάσει πάρα πολλής χρόνος μέχρι να παρουσιαστεί πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επιπλέον, για τα θέματα που έχουν σχέση ε, με συναπόφαση σε δεύτερη ανάγνωση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει να καθορίσουμε μια αυστηρή χρονική περίοδο και αυτή η αυστηρή χρονική περίοδος θα πρέπει να γίνεται σεβαστή απολύτως από τις ε, αρμόδιες επιτροπές ώστε να μπορεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει την άποψή του ε, χωρίς μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με την παρουσίαση της άποψη του Συμβουλίου. Όσον αφορά τώρα το μέγεθος των επιτροπών, το πρόβλημα είναι ότι μπορεί ε, οι δύο κοινέ επιτροπές που ασχολούνται με το θέμα να έχει πολύ περισσότερα μέλη και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ψηφοφορία εάν γίνει μόνο ε, με δόν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποιος περιορισμός και ίσως ε, μία λύση θα ήταν να απαιτείται πλειοψηφία και στις δύο επιτροπές για το θέμα. Ή τέλος πάντων κάποια άλλη λύση. Όπως και να έχει από τώρα μέχρι τις 31 Μαρτίου που έχουμε θέσει ως καταληκτική ημερομηνία για την παρουσίαση τροπολογιών, ε, η ομάδα μου εκ μέρους του κυρίου Ντέβιτ Μάρτιν θα παρουσιάσει σχετικές τροπολογίες για να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε λίγο τη διαδικασία, να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια γρήγορη διαδικασία από πλευράς χρόνων και μπορούμε να έχουμε και ε, κατάλληλες αρμοδιότητες και ψηφοφορίες στις δύο επιτροπές ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον αριθμό των μελών της κάθε επιτροπής. Ο κύριος Χέφνερ. Ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις και σας κύριε Πρόεδρε και για την συζήτηση και επειδή έχουμε χρόνο θα ήθελα να καταθέσω κάποιες σκέψεις, ερωτήματα χωρίς να είναι τελικές κρίσεις. Τα ζητήματα πάνε τώρα στην εξή κατεύθυνση. Εγώ ίδιος δεν είμαι σίγουρος για το εάν ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε τόσο αυστηροί στη ρύθμιση όσο αντιλαμβάνομαι εγώ ότι είναι αυτή η πρόταση. Γιατί υφίσταται ο κίνδυνος, όπως είπατε, αλλά μπορεί να είναι και μια ευκαιρία. Μιλήσαμε για διεπιστημονικότητα. Βλέπουμε πως ε, σε πράγματα τα οποία βεβαίως ε, συνδυάζονται ε, βλέπετε πως οι επιτροπές εργάζονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη και όσον αφορά το, το νομικό τμήμα αλλά και τις πολιτικές θέσεις. Ε, είναι τελείως διαφορετικές οι απόψεις που, στις οποίες καταλήγουν οι επιτροπές, κάτι το οποίο κοστίζει και χρόνο, αλλά θα έπρεπε να είχαμε ίσως ένα ευρύτερο έτσι αποτέλεσμα αν τα εξετάζαμε τα πράγματα από περισσότερες πτυχές και πλευρές και θα γλιτώναμε χρόνο στο τέλος. Ε, είχαμε μια ενδιαφέρουσα εμπειρία παραδείγματο χάρη ε, με την έκθεση που κάναμε για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που συνεργαστήκαμε με τρεις άλλους συναδέλφους από τρεις άλλες επιτροπές και ορισμένες φορές νομίζω πως το να ερχόμαστε σε συνεννόηση με διαφορετικές επιτροπές, με διαφορετική οπτική μπορεί να εξυπηρετήσει νομίζω και το κοινοβούλιο και το τελικό αποτέλεσμα. Και αυτό το έδειξε και η τελική ε, ψηφοφορία, πως ήταν καλό το ότι ξεκινήσαμε με δύο επιτροπές που είχαν διαφορετική οπτική γωνία. Αυτό έτσι απλά ως ερέθισμα για σκέψη. για το ζήτημα το οποίο συζητάμε σήμερα. Δηλαδή μπορεί πάρα πολλές φορές ε, να αποδειχθεί πλεονέκτημα αυτό το οποίο θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί το Κοινοβούλιο. Yeah. Ε, ναι. Και εγώ δεν έχω συγκεκριμένη πρόταση, απλά θα ήθελα να αναφέρω πως πράγματι αυτό το οποίο μόλις ακούστηκε περί κοινών ε, συνεδριάσεων και προεδριών των επιτροπών. Νομίζω πως είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Έχω πει πως και το άρθρο 50 και το άρθρο 51, ειδικά όσον αφορά την Επιτροπή Γιούρι και Ίμκο που κατά κανόνα διαφέρουν, γίνεται όλο και πιο σημαντικό γιατί οι επιτροπές έχουν μια κάποια κοινή αρμοδιότητα και θεματολογία και θα πρέπει να αποφύγουμε το ότι η πολυπληθέστερη επιτροπή απλά να έχει περισσότερες ε, ψήφους και να επιβάλλει την, ε, την άποψή τους. Όχι, θα πρέπει να υπάρχει μια ίση εκπροσώπηση. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω βεβαίως. Ευχαριστώ, κύριος Βίλαντ. Ε, με συγχωρείτε, παίρνω ξανά το λόγο, αλλά άκουσα τους συναδέλφους. Πράγματι, είναι πρόβλημα όταν οι επιτροπές από το μέγεθός τους και μόνο δημιουργούν έτσι σύγχυση. Και βεβαίως όχι όταν δημιουργούνται πλειοψηφίες, αλλά όταν παραμένουν τα ζητήματα επίμεχα. Κοιτάξτε, στην διάσκεψη ΑΚΕ έχουμε την πλειοψηφία και των δύο ε, σωμάτων αλλά αυτό είναι ένα είδος βέτο. Έχουμε και αυτά τα μηχανηματάκια εδώ πέρα μπροστά μας ψηφοφορία, οπότε θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε και να κάνουμε τι όμως, όχι τον αριθμό, αλλά το ποσοστό των ψήφων στην κάθε επιτροπή και μετά να πούμε αυτή είναι η πλειοψηφία και θα έχει λυθεί έτσι το ζήτημα του μεγέθους της κάθε επιτροπής. Λοιπόν, περιμένω τις τροπολογίες σας για να αξιολογήσω και πιο προσεκτικά τις επιφυλάξεις που παρουσιάσατε. Κάποιες διευκρινήσεις όμως ήδη εκ των προτέρων μπορούμε να κάνουμε. Καταρχάς, το θέμα της διακριτικής ευχέρειας. Εμείς ξεκινάμε από το άρθρο 51, το οποίο λέει ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου κανόνα μπορεί να γίνει μόνο όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 41 και του άρθρου 50 και επομένως η διακριτική ευχαίρεια είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που προτείνεται εδώ και η προσπάθεια που κάνουμε είναι ακριβώς να μην το αφήνουμε στη διακριτική ευχαίρεια κανενός διότι τα άρθρα 49 και τα άρθρα 50 είναι πολύ αμφίσιμα. Το άρθρο 50 απλώ παρουσιάζει κάποιε κοινέ αρμοδιότητε. Ε, είτε είναι μεγάλε είτε μικρέ. Εδώ μιλάμε για ε, περιπτώσει τι οποίε έχουν ουσιαστικά σύνδεξη. Είναι τελείω αδύνατο να καθορίσουμε ποιο έχει την αρμοδιότητα για ένα συγκεκριμένο θέμα μεταξύ δύο επιτροπών. Εδώ είναι το θέμα λοιπόν. Ε, θα προσπαθήσω να το τελοποιήσω, αλλά εκτό και αν διαγράψουμε το άρθρο 50, δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε λύση. Αλλά εκεί προκύπτουν άλλε επιπλοκέ. Μπορεί μια μη αρμόδια επιτροπή να αναλάβει ένα θέμα το οποίο μπορεί να μην είναι αρμοδιότητά τη ε, και να μην έχει τη δυνατότητα να επιλύσει ένα ζήτημα. Όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα, το θέμα είναι πολύ σοβαρά. Ε, κάποιος αναφέρθηκε στη διάσκεψη των Προέδρων. Η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών είναι αρμόδια για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να απλουστεύσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη διαδικασία όταν έχουμε κοινέ επιτροπέ που ασχολούνται με το ίδιο θέμα ε, σε σχέση με τη διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης ε, διότι πρέπει να γίνονται σεβαστά και κάποια χρονικά περιθώρια. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια περαιτέρω απλούστευσης, κυρίως για το τελικό στάδιο, την εκτελεστική διαδικασία. Και εκεί έχουμε προτείνει να μην είναι οι κοινέ επιτροπές ε, οι οποίες ε, υποχρεωτικά θα πρέπει να παρακολουθούν την εκτέλεση, αλλά να μπορεί να αναλάβει το καθήκον αυτό μόνο μια επιτροπή. Ε, ποιο αποφασίζει όμω ποια θα είναι η αρμόδια επιτροπή, ποιο αποφασίζει ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού. Αν εμεί χάσουμε χρόνο σε αυτή τη διαδικασία, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Επομένω, χρειάζεται ε, ένα όργανο, κάποιο, ίσω και ο πρόεδρο, και να λύσει το θέμα εκεί. Αλλά ε, θα σας παρουσιάσω κάποιες τροπολογίες, θα το σκεφτείτε κι εσεί μαζί με μένα και θα βρούμε την καταλληλότερη λύση. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσει, νομίζω ότι μπορούμε να ε, θεωρήσουμε ότι τελειώνει η συνεδρία τη Επιτροπή και θα ξεκινήσει εντό ολίγου η συνεδρία των συντονιστών. Ευχαριστώ λοιπόν ε, τα μέλη τη Επιτροπή σε αύριο.